Καλημέρα συνάδελφοι. Κάποιες ανακοινώσεις να κάνω όσον αφορά τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές χθες. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την έκθεση την προ... για την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αναστέλει προς όνομα της αυτόνομους τελωνιακούς δασμούς για κάποια βιομηχανικά προϊόντα των αυτονόμων περιοχών Μαδέρας και Αζωρών αυτό είναι κάτι που αναλαμβάνει ο Πρόεδρος. Δεύτερον, οι γνωμοδοτήσεις όσον αφορά την πρώτη κανονισμού του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό που καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα για τη γεωργία στις υπεραπομακρυσμένες περιοχές της ενώσεως ανατίθεται στο ΕΛΚ, στην ομάδα του ΕΛΚ. Δεύτερον, η γνωμοδότηση Ρέτζι... όσον αφορά την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2008, κεφάλαιο 3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανατίθεται στην ομάδα του ΕΛΚ. Το σχέδιο εκθέσεως για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ετήσια έκθεση 2008, Τάμας Ντόιτς του ΕΛΚ αναλαμβάνει Σχέδιο εκθέσεως για τα οικονομικά συμφέροντα της κοινότητα και καταπολέμηση των απατών ετήσια έκθεση του 2008 αναλαμβάνεται από το ΕΛΚ. Α, συγγνώμη, λέει ο πρόεδρος. Εντάξει, στο ΕΛΚ πάει. Σχέδιο εκθέσεων αφορά τις νέες εξελίξεις όσον αφορά τις ε, κρατικές προμήθειες. Χάιντε Ρούλε της ομάδας ERC. Προθεσμία. Α, όσον αφορά την ακρόαση του νέου επιτρόπου, προθεσμία για τοποποίηση του παρατήματος σημείου 5 του κοινού σχεδίου ερωτηματολογίου είναι 5η 5 Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Αντιπροσωπείες. Οι ακόλουθες αντιπροσωπείες για το 2010 έχουν συμφωνηθεί. Γαλλία ΕΛΚ, Γερμανία Σαντί, Βραζιλία ΕΛΚ και ΓΚΟΕ. Δημόσια Κροασία. Έχουμε συμφωνήσει για ακροάσεις που ενεκρίθησαν το 2000 για το 2010. Πρώτα απ' όλα προς μία επίδοση με στόχο ότι αποτελέσματα όσον αφορά την πολιτική συνοχής ΕΛΚ. Πολιτικές αστικής ανάπτυξης Πράσινη, άντε και ECR ε, έχουν κάνει την πρόταση. Άτυπη ομάδα εργασίας που απαρτίζεται από ένα άτομο αναπολιτική ομάδα, ένα ε, αναπληρωματικό μέλος από την Άντε θα δημιουργηθεί, θα προετοιμάζει το έργο, οι αποφάσεις θα θα λαμβάνονται στην Επιτροπή Ρέτζη θα κοινοποιούν οι ομάδες τα μέλη τους, τους εκπροσώπους τους στη γραμματεία, το ταχύτερο δυνατόν να σκηνοποιήσουν τα μέλη που θέλουν να στείλουν εκεί. Τόσο αναφορά αφορά τι μελέτε, οι ομάδες μπορούν να στείλουν προτάσει στη γραμματεία μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Απόφαση θα ληφθεί το Δεκέμβριο, το αργότερο. Ας πάμε λοιπόν στην ε, ημερήσια διάταξή μας. Συγγνώμη Πρόεδρε, ίσως να μην κατάλαβα κάτι. Η συγητής για τη γνωμοδότηση της έκθεσης για την Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων για την ετήσια έκθεση του 2008 αναλαμβάνεται από το SED. Όχι, SND. Προχωράμε στο πρόγραμμα. Στο σημείο, το σημείο 7 θα συζητηθεί αν έχουμε χρόνο μετά την ψηφοφορία. Κυρία Κέλλη. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλημέρα. Να υπογραμμίσω ότι η αντιπροσωπεία που θα πάει στη Γαλλία παρουσιάζεται και κάποια πρόταση σχετικά από το ΕΛΚ όσον αφορά το θέμα των ερευνών, της έρευνας και το δεύτερο τμήμα το παρουσιάσουν οι πράσινοι όσον αφορά τα προάστια. Αυτό προς ενημέρωσή σας. Όσον αφορά τι αντιπροσωπείε, Γαλλία μετά πρόταση του ΕΛΚ να συνδυαστεί δυνατόν με τους πρασίνους και την πρότασή της Άλτε Συμφωνείτε, Λαμπέρτ Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Σωστή είναι η ανάθεση των εισηγητών στους το των θεμάτων. Θα ήθελα να τα δω επί χάρτου για να είμαι βέβαιος ότι όλα έχουν γίνει σωστά. Θέλω κείμενο. Δεύτερον, σωστά τα της αντιπροσωπείας. Το ΕΛΚ πρότεινε κάποια πράγματα. Πρέπει να συζητήσουν οι συντονιστές και στο τέλος καταλήξαμε σε συμπεράσματα. Το ΕΛΚ πρότεινε... Το ΕΛΚ είχε προτείνει για τη Βραζιλία. Έγινε συζήτηση μεταξύ συντονιστών και είπαμε αυτές είναι οι χώρες έγιναν παρατηρήσεις για την Γαλλία, αλλά δεν είναι κάτι πολιτικό. Είναι απόφαση των συντονιστών των επιτροπών που ελήφθη. Ήταν θέμα συγκεκριμένη πολιτικής ομάδας. Λοιπόν, να προχωρήσουμε, λέει ο Πρόεδρος, να προβούμε στην ψηφοφορία. Επιθυμώ να τονίσω και πάλι ότι θα επεξεργαστούμε μαζί την ατζέντα αυτής της αντιπροσωπεία και ότι από κοινού όλα αυτά αποφασίστηκαν στη συνάντηση των συντονιστών. Βλέπω ότι συμφωνεί και η Κωνσταντσε Κρέλ νεύοντα καταφατικά. shall we go ε, ας, Ας προχωρήσουμε μάλλον στην ημερήσια διάταξη. Όπως σας είπα πριν, το σημείο 7 θα αναβληθεί. Θα συζητηθεί μετά την ψηφοφορία. At the would you please check your electronic... Ελέγξτε παρακαλώ τα μηχανήματά σας, τις κάρτες σας, να δείτε αν λειτουργούν μηχανήματα για την ψηφοφορία. My does work. So we open the vote. If everybody has put the, the, the card, we open. If everybody has inserted the card. Λοιπόν, έχετε όλοι τις κάρτες σας. Ωραία, μπορεί να ξεκινήσουμε την ε, ψηφοφορία. Ξεκινάμε.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 So it seems to be everything is okay. Όλα πηγαίνουν καλά φαίνεται. Somebody has a problem. Sorry? Ah, the voting list, the voting. Okay. Yes, we, we wait, we wait a minute until. Να περιμένουμε ένα λεπτό μέχρι ότου διανεμηθεί ο κατάλογο ε, ψηφοφορία από το ΕΛΚ. Yes, please. Yes, please. Ε, καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Από την Ελλάδα είμαι, είμαι νέος βουλευτής Δυστυχώ δεν έχω κάρτα ηλεκτρονική, αλλά θα ήθελα να συμμετέχω στην ψηφοφορία. Αν μπορείτε να με διευκολύνετε. Μπορείτε να ψηφίζετε με το χέρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνω είναι θετική ψήφο, κάτω είναι αρνητική και οριζόντιο είναι εποχή. Πάνω θετική, κάτω αρνητική, οριζόντιο ε, μηδέν. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ και καλώ ορίσατε. Να είστε καλά. Uh, we only, we only need the, the when, there is a, a problem, eh, when I don't see clear, Okay. okay, we can start ξεκινήσουμε. Επιλεξιμότητα όσον αφορά των παρεμβάσεων για τη στέγαση υπέρ των περιθεροποιημένων κοινοτήτων. Ξεκινάμε τροπολογία 12 με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Οι 13, οι 14 και οι 15 καταπίπτουν συνεπώς. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία. Η τροπολογία 3 καταπίπτει. Απορρίπτεται, λέει ο πρόεδρος. Ποιος είναι υπέρ για την 3. Ποιος είναι υπέρ της 3. Κατά της 3. Αποχές. εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται οι τροπολογίες 4 και 5 θα ψηφιστούν ομού διότι είναι ταυτόσιμες ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αποχέ ο πρόεδρος εγκρίνεται. 7 καταπίπτει. 8 καταπίπτει. 1 Ψηφίζουμε την τροπολογία 8, υπέρ της 8 κατά αποχές απορρίπτεται. 1. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. if is adopted. Καταπίπτει εάν υιοθετηθεί η 8. Αν εγκριθεί η 8. Πρέπει να ψηφίσουμε συνεπώ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά ηλεκτρονικά Ξεκινάμε. Open the vote. Open the vote, please. Αρχίζει η ψηφοφορία. Τώρα πέρα στις ψηφοφορίες. Λειτουργεί. 38 εψήφισαν, 34 υπέρ, 3 κατά, μια αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν το σχέδιο εκθέσεως και συγχαρητήρια στον εισηγητή. Now we proceed. Θα προχωρήσουμε στο 9 γνωμοδότηση για το σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού. Τροπολογία υπαριθμών 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Υπαριθμών 6. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 εδώ ζητείται ψηφοφορία κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ όχι δεν είναι έτσι Ναι, ναι, μάλιστα. Είναι η ψηφοφορία κατά τμήματα. Λοιπόν, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτό. Α, απορρίπτεται, απορρίπτεται, συγγνώμη. Εκπίπτει η, ε, η 7. Τώρα, τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Αυτή εγκρίνεται. 8. Εδώ ζητείτε πάλι ψηφοφορία κατά τμήματα. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Α, το επόμενο εκπίπτει το 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και αυτή 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται υπαριθμών 9 και 27 μαζί διότι είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Όπως βλέπετε. Πρέπει να ψηφιστεί λοιπόν 28 υπέρ. Κατά. Αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. μόνο 10 υπέρ κατά εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31. Α, έχει αποσυρθεί. Υπάρχει μόνο ένα. Υπέρ, κατά, αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση αρχίζει η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται υπαριθμών 12 υπέρ κατά εγκρίνεται 13 με προφορική τροπολογία. Όπως βλέπετε στην λίστα σας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, Α, εγκρίνεται. 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Υπάρχουν 2 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Καλώς. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη λοιπόν. Υπαριθμούν 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκπίπτει υπαριθμών 3. 4. Υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση αρχίζει η ψηφοφορία κλείνει η ψηφοφορία εγκρίνεται τελική ψηφοφορία γίνεται ηλεκτρονικά αρχίζει ακούσατε όλοι. Εγκρίνεται. Με 38 ψήφους υπέρ, μία κατά και δύο αποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Α, θες να δώσω λόγο στον κύριο Λόφα, αλλά είναι απόν.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 So, dear colleagues, we will start. Αγαπητοί. φίλοι, σε ένα λεπτό θα αρχίσουμε. So, shall we start, dear colleagues? Yes. Έχετε όλοι το κείμενο της ε, παρουσίασης PowerPoint. Φαίνεται πως όλοι την έχουν. Οι διερμηνείς δεν την έχουν. Πρώτα απευθύνω το καλωσορίσατε στον κύριο Μέλμπι και του δίδω το λόγο για να κάνει την παρουσίαση. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρόσκληση να προσέλθω εδώ στην απολύτως νέα Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης για να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα ΕΣΠΟΝ. Θα σας πω με λίγα λόγια τι γίνεται στο πρόγραμμα. για την χορήγηση στοιχείων και δεδομένων για την ανάπτυξη Τη δυναμικότητα των περιφερειών μέσα στο ευρωπαϊκό, στην ευρωπαϊκή επικράτεια. Θα σα πω λίγα λόγια πρώτα για την αποστολή μας, καθώς και για τι προτεραιότητε του προγράμματο και για την πρόοδο που έχουμε επιτελέσει άχρη τούδε. Μετά θα σας πω λίγα ε, λόγια για τα παραδείγματα για, τις, ε, για το output του προγράμματος του ΕΣΠΟΝ και εν τέλει κάποιες ας πούμε σκέψεις ως συμπεράσματα για και την ανταλλαγή ε, δεδομένων από την ΕΣΠΟΝ προς εσάς και σχετικά με τα όσα ήδη έχουν συζητηθεί για το πρόγραμμα του ΕΣΠΟΝ. Πρώτα, ε, χρηματοδοτούμεθα από τα τα ταμεία μέσα στη, στον στόχο της ε, Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Territorial Cooperation και έχουμε στοιχεία και δεδομένα για τις προοπτικές, τις τάσεις, τις επιπτώσεις της άσκησης των πολιτικών που επηρεάζουν την, τις περιφέρειες καθώς και την ανάπτυξή τους. Και η αποστολή μας είναι να παράγουμε συγκρίσιμες πληροφορίες και ιδιαίτερα να δείχνουμε πού βρίσκεται το δυναμικό ανάπτυξης των διαφόρων μερών της Ευρώπης. Έχουμε έναν προϋπολογισμό περίπου 47 εκατομμυρίων ευρώ από τα οποία το 75% προέρχεται από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα υπόλοιπα χρηματοδοτούνται από τις χώρες μέλη. Με συνολικά 31 χώρες, 31 χώρες ε, μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, δηλαδή είναι και τέσσερις χώρες εταίροι. Είμαστε το πρόγραμμα που έχει τις περισσότερες ε, χώρες ε, που αναμειγνύονται. Οι χώρες όπως βλέπετε είναι η Ελβετία, η Νορβηγία, το Λίχτενστάιν και η Ισλανδία. Εφαρμόζουμε πέντε προτεραιότητες. Η πρώτη και πιο σημαντική είναι η εφαρμοσμένη έρευνα για να κατανοήσουμε καλύτερα την δυναμική μέσα στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Έχουμε έξι ε, προγράμματα, project, τα οποία προχωρούν. Θα δείτε ότι ρίχνουμε ιδιαίτερο βάρος στα αστικά κέντρα και τις πόλεις, ιδιαίτερα στη λειτουργικότητα των περιοχών αυτών που θεωρούμε ότι είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για τον καθορισμό και την ανάπτυξη των στρατηγικών για το μέλλον, εξετάζουμε τις δυνατότητες ευκαιρίες ανάπτυξης σε διάφορες περιοχές της Υπέθρου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Υπέθρος στην ε, Ευρώπη είναι πάρα πολύ διαφορετική, δημογραφικά και μεταναστευτικά ρεύματα, Επίσης, ενέργεια, επίσης, καθώς και αύξηση των τιμών της ενέργειας, που εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο μας απασχόλησε πάρα πολύ, οι επιπτώσεις δηλαδή στις περιφερειακές οικονομίες αυτών των ε, διακυμάνσεων των τιμών της ενέργειας, κάνουμε και ένα territorial impact assessment το οποίο η πολιτική πλευρά μας το ζητά επίμονα εδώ και καιρό και τέλος το θέμα της αλλαγής του κλίματος που επίσης έχει περιληφθεί στο πρόγραμμα του ΕΣΠΟΝ. Προετοιμάζουμε και 11 νέα project τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν ε, βγει σε ανοιχτή ε, διαδικασία πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος και θα δείτε εδώ τους βασικούς τίτλους που έχουμε επιλέξει και έχουν επιλέξει δηλαδή όλες οι αναμειγνιόμενες χώρες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ε, συμβουλευτική, συμβουλευτικό όργανο στην περίπτωσή μας με θέματα τα οποία πρόκειται να ανατεθούν πλέον με συμβάσεις τέλη του χρόνου και αρχές του καινούριου χρόνου και τα αποτελέσματα θα τα έχετε και εσείς διαθέσιμα για το έργο σας. Θα δείτε ορισμένα από αυτά όπως η ελκυστικότητα των περιφερειών και ε, πόλεων, ε, η τρόπη όπου χρησιμοποιείται, χρήσης γης δηλαδή στην Ευρώπη, η περιφερειακή, εδαφική συνεργασία, η δημιουργία νέων και ίσως μεγαλύτερων περιφερειών όπως αυτήν της ε, Βαλτικής, η προσβασιμότητα των ε, περιφερειών που έχει επίσης πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει και στο περιφερειακό ε, επίπεδο αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο θα σας δείξω και χάρτες σχετικά μετά από λίγο δευτερεύοντες πόλη ανάπτυξης που επίσης είναι σημαντική στην περιφερειακή ανάπτυξη. Θα εξετάσουμε και τα διάφορα εδάφη τα οποία έχουν ε, ζητηθεί μέσα στην ε, συνθήκη η οποία βέβαια υπεγράφει τέλος και από την τσεχική δημοκρατία χθε και πρόκειται να τεθεί σε ισχύ θα θυμάστε ότι υπάρχουν ορισμένα εδάφη territories που έχουν σχέση με την ε, εδαφική συνοχή, για παράδειγμα ορεινές περιοχές, νησιωτικές περιοχές και ούτω Θα προσπαθήσουμε να ε, δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο πληροφόρησης και γνώσης για τις ε, περιοχές αυτές. Επίσης η οικονομία της πληροφορίας, οι υπηρετικές εδαφικές δομές σε σύγκριση μεταξύ Ευρώπης και του κόσμου σύγκριση δηλαδή της Ευρωπαϊκής Υπήρου με τον υπόλοιπο κόσμο έχουμε ήδη ένα project το οποίο έχει, αναφέρεται στην Ευρώπη και στον κόσμο και εδώ πρόκειται για μια προσπάθεια εμβάθυνσης των όσων έχουμε ήδη ξεκινήσει. Υπηρεσίε υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος, κοινή ωφέλεια δηλαδή, οι ευρωπαϊκές θάλασσε δραστηριότητε δηλαδή και ε, πήγες αλλά και ε, μια δηλαδή συνέχεια του Territorial Impact Assessment, να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους να κάνουμε μια σάρωση, ένα σκάνινγκ των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σχέση με το θέμα της ε, εδαφικής ανάλυσης. Και όλα αυτά καθορίζονται από τις χώρες μέλη και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από τις χώρες εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΟΝ. Άρα πρόκειται για μια εκ των άνω ε, ανάλυση του προγράμματος. Έχουμε όμως και ένα στοιχείο εκ των κάτω, όπου το βασικό που μας απασχολεί είναι να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που διαθέτουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο σε συγκεκριμένα project, πάλι μαζί με τους ενδιαφερόμενους. Εδώ ζητούμε από τους ίδιους ενδιαφερόμενους να έλθουν από την ρίζα, δηλαδή να μας προσφέρουν ιδέες για θέματα όπου θέλουν να βάλουν μια ευρωπαϊκή διάσταση για το μέλλον. Έχουμε ορισμένα ε, προγράμματα, ορισμένα project τα οποία ήδη ξεκινούν με διάφορους, με διάφορους συσχετισμούς εταίρων. Βλέπετε και στην διαφάνεια που δείχνω τώρα ότι δίνεται ιδιαίτερη, ε, ιδιαίτερη σημασία σε, ε, στις οικονομίες διαφόρων μεγάλων αστικών κέντρων όπως Μάντσεστερ, Βαρκελόνης, Δουβλίνου και Λιών. Ιδιαίτερα εξετάζουμε επίσης το θέμα των νησιών όπου εδώ συμμετέχει το Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδος μαζί με άλλους εννέα ενδιαφερόμενους. Το τρίτο είναι επίσης πολύ σημαντικό, η προσπάθεια να φτιάξουμε πολυκεντρικά μητροπολιτικά κέντρα, ε, οι περιφέρειες οι οποίες θα συνδυαστούν με άλλες πολυκεντρικές δομές που έχουν και διαμεθοριακές συνεργασίες και γύρω από το Λουξεμβούργο αλλά και προς νότον της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ελβετίας. Σε άλλο project προσπαθούμε να κατανοήσουμε γιατί ορισμένες από τις ε, περιφέρειες της σύγκλησης είναι επιτυχημένες και άλλες όχι. Έχουμε και τα διάφορα σενάρια τα οποία μπορούν ενδεχομένω να εφαρμόζονται και σε μικρότερο γεωγραφικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα βλέπετε εδώ περιφέρειες τη Βαρκελόνη, του Τουρίνου και του Ερώ και την ποικιλότητα των ε, ε, περιφερειών, πάλι ε, με συμμετοχή ορισμένων υπουργείων και τι χώρε τις βλέπετε εκεί. Δηλαδή, ζητούμε να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τα κάτω και να προσφέρουμε στους ενδιαφερόμενους στοχευμένη ανάλυση, να τους ε, προσφέρουμε δηλαδή τη δυνατότητα να βάλουν την ευρωπαϊκή διάσταση σε αυτά που τους, ενδιαφέρει, που τους ενδιαφέρουν και αυτά βέβαια χρηματοδοτούνται πλήρως από το πρόγραμμα ESPOL. Έχουμε και ορισμένες νέες στοχευμένες αναλύσεις οι οποίες πρόκειται να ε, δημοσιευτούν και για την ώρα έχουμε ζητήσει πάλι νέα έκφραση ενδιαφέροντος και φαίνεται πως αυτά τα project προκαλούν ευρύ ενδιαφέρον στις περιφέρειες και πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Αναμένουμε λοιπόν σημαντικό αριθμό αιτήσεων σχετικά. Βέβαια, παίζουμε και τον ρόλο μας ενός επιστημονικού προγράμματος δηλαδή, διότι επιστήμονες είναι αυτοί που κάνουν τις αναλύσεις, πρόκειται για καθηγητές πανεπιστημίων σε ολόκληρη την Ευρώπη που συνδυάζονται και με ε, εταίρους από τον ιδιωτικό τομέα διεξάγουν αυτή την έρευνα και την ανάλυση λοιπόν για λογαριασμό μας. Άρα δημιουργούμε, παράγουμε και μια επιστημονική πλατφόρμα ώστε σιγά σιγά να δημιουργήσουμε όπως είπα μια επιστημονική πλατφόρμα για ένα είδος territorial science στην Ευρώπη. Και ένα από τα κύρια θέματα είναι βέβαια και η τράπεζα δεδομένων του ΕΣΠΑΝ, όπου περιλαμβάνουμε πολλούς νέους δείκτες και πολύ περισσότερους δείκτες από αυτούς που μπορεί να προσφέρει η Ευρωστάτ. Και ε, τους, ε, κάνουμε, τους ε, διαθέτουμε αυτούς τους δείκτες και μέσω της ιστοσελίδας μας και με άλλους τρόπους που υποστηρίζουν την επιστημονική αυτή προσέγγιση ώστε να δημιουργηθεί ένας ευρωπαϊκός ερευνητικός χώρος για την Territorial Science. Υπάρχουν και αυτοί οι εδαφικοί δείκτες, territorial indicators. Αυτή τη στιγμή αναζητούμε τι μπορούμε να περιλάβουμε εκεί. Και όπως είπα, αυτή η διαδικασία πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι ανοιχτή μέχρι τις 11 Νοεμβρίου. Έχουμε και σημαντική κεφαλαιοποίηση ε, κάνουμε και πολλές δημοσιεύσεις. Δεν έφερα μαζί μου ε, σήμερα ε, δημοσιεύσεις. Έχουμε όμως έναν αριθμό δημοσιεύσεων. Κάνουμε και territorial observations με σύντομα κείμενα περίπου 20 σελίδων με χάρτες όλες που έχουν το στόχο να ενημερώσουν ειδικές ομάδες όπως για παράδειγμα την Επιτροπή σας και αν ενδιαφέρεστε μπορώ να σας διαβιβάσω σημαντικό αριθμό τέτοιων εγγράφων. Κάνουμε και συνοπτικέ εκθέσει όπου προσπαθούμε μέσα σε μια εκατοστή σελίδων περίπου να δώσουμε τι πληροφορίε σε αυτού οι οποίοι λαμβάνουν τελικά τι πολιτικέ αποφάσει σχετικά με εξελίξει και με τα δεδομένα τα οποία έχουν παραχθεί από την έρευνά μα. Εν τέλει υπάρχει και μια αποκεντρωμένη διάρθρωση του προγράμματος του ΕΣΠΟΝ. Υπάρχουν δηλαδή τα contact points σε κάθε χώρα και η μόνη χώρα που δεν έχει τέτοιο contact point είναι το Liechtenstein, το οποίο όμως καλύπτεται από το contact point της Ελβετίας. Τα contact point του ESPON έχουν ως στόχο να προσπαθήσουν ε, να συμβάλλουν σε μια κεφαλαιοποίηση και στο ε, υπερεθνικό επίπεδο. Συνοψίζοντας αυτήν την σύντομη ενημέρωση σχετικά με το τι είναι το πρόγραμμά μας, θα πω μόνο ότι βρισκόμαστε περίπου στα μισά του δρόμου. Του χρόνου το καλοκαίρι θα έχουμε προχωρήσει περισσότερο. Προσπάθησα να σας ε, δείξω με σύντομο τρόπο τις διάφορες δραστηριότητες ε, που έχουμε ξεκινήσει από τότε που αρχίσαμε το πρόγραμμα αυτό μέχρι το 2013 δηλαδή για να ε, σας δώσω όπως είπα μια σύντομη ενημέρωση ελπίζω ενδιαφέρουσα κάνουμε και ένα screening των ενδιαφερόντων των διαφόρων ε, ε, ομάδων, των ενδιαφερομένων δηλαδή, και ένα δεύτερο screening το οποίο θα γίνει του χρόνου και ελπίζω να, ότι θα συμφωνήσετε να περιληφθούν και ορισμένα μέλη της ίδιας της Επιτροπής σας, ώστε να έχουμε ε, και μια εισρωή των πολιτικών ενδιαφερόντων που έχετε εσείς περί τα μέσα του επόμενου έτους μάλλον θα σας προσεγγίσουμε ε, για το θέμα αυτό. Μίλησα πολύ για το τι είναι το ΕΣΠΟΝ. Ήθελα όμως να σας δείξω λίγο και τι είναι και δεν μπορεί παρά να είναι ένα τμήμα μόνο ε, των ε, όσων παράγουμε, των εκρών μας δηλαδή. Σας δείχνω αυτή τη διαφάνεια που δείχνει την Ευρώπη αριστερά Εάν δώσετε στην κάθε περιφέρεια ένα αναλογικό βάρος σε σχέση με τον πληθυσμό της και δεξιά αν δώσετε το μέγεθος ανάλογα με την συμμετοχή της στο κατακεφαλήν εισόδημα. Αν υπήρχαν οι ίδιες συνθήκες για όλους θα βλέπατε τον συνήθι χάρτη της Ευρώπης. Βλέπετε λοιπόν με τον τρόπο αυτό τις ανισότητες που ε, προκύπτουν μέσα στο ε, ευρωπαϊκό έδαφος. Υπάρχουν, υπάρχει ένας αριθμός προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και θα τις γνωρίζετε τις περισσότερες. Όλες αυτές οι προκλήσεις έχουν και κάποιες α, συγκεκριμένες επιπτώσεις στις διάφορες περιφέρειες, στα διάφορα τμήματα της Ευρώπης, στις διάφορες πόλεις. Βεβαίως η οικονομική ανάπτυξη και η ύφεση την οποία βρισκόμαστε. Ίσως υπάρχουν κάποια σημάδια πράγματι ότι αρχίζουμε να μπαίνουμε σε μια θετική πορεία αλλά σίγουρα θα υπάρξουν κοινωνικές επιπτώσεις και του χρόνου για τις ε, περιφέρειες οι οποίες ε, πλήττονται με αυθαίρετο τρόπο βέβαια από τα κλεισίματα επιχειρήσεων κλπ. Το κύριο μήνυμα εδώ είναι ότι βρισκόμαστε σε μια φάση επιταχυνόμενης παγκοσμιοποίησης και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη από κάθε άποψη. Νομίζω λοιπόν ότι θα δούμε την ασιατική οικονομία να παίζει κυρίαρχο ρόλο στον κόσμο και μία από τις καταστάσεις που αντιμετωπίζει η περιφερειακή ανάπτυξη είναι ότι δεν μπορείς πλέον να εξετάζεις μόνο τον εαυτό σου ή μόνο τους άμεσους γειτονές σου. Πρέπει να περιλάβεις στις σκέψεις και στο σχεδιασμό σου ευρύτερα εδαφικά πλαίσια ώστε να μπορέσει η Ευρώπη να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του ενεργητικού που διαθέτει δηλαδή και την σημαντική περιφερειακή ποικιλότητα. Έχουμε και το θέμα της αλλαγής του κλίματος που επίση παίζει σημαντικό ρόλο. Νομίζω η όλη προσέγγιση στην αλλαγή του κλίματος, για παράδειγμα που ενδέχεται να, να, να ανοίγει και νέες δυνατότητες ανάπτυξης σε ορισμένες περιφέρειες της Ευρώπης, δηλαδή η κρίση δεν πρέπει να εξετάζεται μόνο από τις ε, αρνητικές πλευρές της, αλλά και ως άνοιγμα νέων ευκαιριών. Οι δημογραφικές αλλαγές συνεχίζονται. Έχω και ορισμένες ε, διαφάνειες που θα σας τις δείξω σε λίγο. Η πρόκληση το, της ενέργειας, σας τα είπα πριν από λίγο, η αύξηση των μεταφορών θα τα δούμε και στα επόμενα δέκα χρόνια και βέβαια και η γεωγραφική ολοκλήρωση με την έννοια της παραπέρα διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή μας απασχολεί. Ένας αριθμός χαρτών τώρα που δείχνει την δημογραφική εξέλιξη ε, και που είναι ένα μέρος του σενάριου που έχουμε φτάσει, που έχουμε φτιάξει και που είναι ένα σταθερό, μια σταθερά του σενάριου αυτού. Βλέπετε εδώ πώς θα αντιμετωπίσουν οι ευρωπαϊκές περιφέρειες μια, μέσα, μια μέση ηλικία 50 ετών στις πιο σκούρες περιοχές και πώς κατανέμονται μέσα στην Ευρώπη. Εάν δείτε τώρα την πίεση ε, από τη μετανάστευση, θα δείτε ότι η μεγαλύτερη αύξηση ε, πληθυσμού είναι στις ε, βόρειο-αφρικανικές χώρες, νότια της Ευρώπης δηλαδή, και πρέπει να αναμένετε ότι η πίεση την οποία ήδη δεχόμαστε θα αυξηθεί ή θα, ή θα συνεχιστεί πάντως. Έχουμε και ένα project που έχουμε αρχίσει τώρα να δούμε ποια είναι τα μέρη εκείνα τα οποία <clears throat> κυρίως προωθούν την ε, οικονομία στην Ευρώπη θα δείτε ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός συγκέντρωσης των δραστηριοτήτων. Παρακαλώ κάντε ένα κλικ ακόμη. Θα δείτε μέσα σε αυτό το πεντάγωνο, ελπίζω ότι το βλέπετε πάνω στο χάρτη, ότι εκεί έχουμε περίπου παραγωγή του μισού ΑΕΠ της Ευρώπης. Έχουμε περίπου 30% των Ευρωπαίων πολιτών σε ένα περίπου 15% του ευρωπαϊκού εδάφους και αυτοί παράγουν το μισό, όπως είπα, εισόδημα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ συγκεντρωμένος ο τρόπος, συγκεντρωτικός μάλλον ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το εδαφός μας. Υπάρχουν πολλές μεγάλες μητροπόλεις, οι οποίες αναπτύσσονται με ταχύτατο ρυθμό. Βλέπετε με το κόκκινο χρώμα στον χάρτη ότι οι νέες χώρες μέλη προς Ανατολάς αλλά και πιο περιφερειακά μέρη της Ευρώπης, ας το πούμε έτσι, έχουν την μεγαλύτερη αύξηση του ρυθμού ε, ανάπτυξης του ΑΕΠ. Υπάρχουν λοιπόν κάποια σημάδια μιας καλύτερης ισορροπίας και μιας καλύτερης ανάπτυξης μέσα στην Ευρώπη. Τώρα, η στρατηγική, η στρατηγική της Λισαβόνας και οι σχετικοί δείκτες. Και εδώ ε, έχουμε φτιάξει ένα χάρτη πριν από την, δείχνει την κατάσταση πριν από την ύφεση. Βλέπετε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι διάφορες περιφέρειες ε, στην Ευρώπη για να συμβάλλουν στις, ε, στους στόχους μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης βασισμένη στη γνώση. Το μήνυμα εδώ είναι ότι ορισμένες περιφέρειες ίσως να μην πρέπει να ακολουθήσουν μοναχά το δρόμο της ε, κοινωνίας της γνώσης και προφορίας, αλλά και άλλους. Τώρα, η προσβασιμότητα. 7 από 10 περιφέρειες της Ευρώπης έχουν θετικό ΑΕΠ. Θετική προσβασιμότητα, δηλαδή πάνω από το μεσόωρο. Αυτό εννοούμε. Υπάρχει λοιπόν ένα συσχετισμός μεταξύ των δύο αυτών παραγόντων. Βλέπετε εδώ την πολυτροπική ε, προσβασιμότητα, accessibility. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, τι, ποιο αριθμό προσώπων μπορείς, ε, να, είσαι, μπορείς να έχεις πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Βλέπετε λοιπόν εδώ με το multi-model, το πολύτροπο δηλαδή τρόπο μεταφορών που σημαίνει και δρόμο και ε, σιδηρόδρομο και ούτε καθεξής και βλέπετε και μόνο για τους δρόμους πολύ πιο συγκεντρωτικό συγκεντρωτική την εικόνα. Βελτιωμένη προσβασιμότητα δηλαδή, κυρίως προς Ανατολάς, που σημαίνει ότι πολλές από τις χώρες μέλη εκεί έχουν δώσει προτεραιότητα στην κατασκευή έργων υποδομής των αυτοκινητοδρόμων. Εάν πάρετε τώρα τον σιδηρόδρομο, βλέπετε λίγο διαφορετική εικόνα. Εδώ όμως το βάρος δίνεται κυρίως, οι πιο σκούρες περιοχές είναι στην Δύση, διότι έχουν γίνει πιο σημαντικέ επενδύσει εκεί σε τρένα μεγάλη ταχύτητα κλπ. Σε ό,τι αφορά τώρα τι αεροπορικέ μεταφορέ, θα δείτε πολύ πιο πολυκεντρική εικόνα, η οποία μάλιστα έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια μετά από την απελευθέρωση των ε, εναέριων μεταφορών. Και πολλές από τις περιοχές αυτές έχουν γίνει και ανταγωνιστικές, ώστε έχουν πρόσβαση και σε πολλά μέρη της Ευρώπης και εκτός των κέντρων. Και βλέπετε ήδη και από τούτον εδώ τον χάρτη που δείχνει τις τάσεις μεταξύ 2001 και 2006 για τις αεροπορικές μεταφορές, κυρίως στις ανατολικές χώρες είναι αυτές που έχουν υποφεληθεί περισσότερο από την αύξηση της προσβασιμότητας από τον αέρα. Εξετάζουμε επίσης και θέματα που έχουν σχέση με την αλλαγή του κλίματος και έχουμε κάνει και χάρτες της εμφάνισης και επανεμφάνισης 11 διαφορετικών ειδών κινδύνων. Μπορεί να αναλυθεί ο χάρτης αυτός σε τέσσερις χάρτες όπως εξής. Για παράδειγμα, οι επανεμφανίσεις πλημμυρών, πυρκαγιών δασών και ούτε καθεξής. Δείχνουμε εδώ δηλαδή ποιους κινδύνους αντιμετωπίζουν οι χώρες μέλη και ποιοι θα έπρεπε να τις απασχολούν εφόσον έχουν κάποιες σχετικές αμφιβολίες. Το κύριο μήνυμα εδώ είναι να πούμε ότι αυτό που πρέπει να αναμένουμε είναι ότι οι αλλαγές κλίματος θα αλλάξουν την πυκνότητα αυτών, την συχνότητα αυτών των ε, ε, φαινομένων καθώς και την έκτασή τους. Αυτό θα πρέπει να αναμένεται και να ληφθεί υπόψη για το μέλλον. Τελευταίε δύο διαφάνειες. Ευρώπη και κόσμος. Δεν μπόρεσα να αντισταθώ στον πειρασμό να σας δείξω μια-δυο διαφάνειες που να δείχνουν ότι βέβαια για την Ευρώπη πρέπει να σκεφτούμε την θέση μας μέσα στον κόσμο. Και γι' αυτό κάνουμε και έχουμε και ένα project εφαρμοσμένης έρευνας εδώ. Θα δείτε το βάρος του ευρωπαϊκού πληθυσμού, ότι έχει δηλαδή μειωθεί μέσα στα τελευταία 50 χρόνια η σχετική δηλαδή ε, βαρύτητα του πληθυσμού αναλογικά με τον υπόλοιπο κόσμο. Και το ίδιο θα δείτε στην επόμενη ε, διαφάνεια σχετικά με το καθόριστο, με το καθόριστο εθνικό προϊόν. Ίσως λοιπόν πρέπει να δούμε πιο σφαιρικά την Ευρώπη και να δούμε η περιφερειακή ανάπτυξη πώς μπορεί να συμβάλλει στην ε, ανάπτυξη γενικότερα, δηλαδή στη γενικότερη, συνολικότερη ανάπτυξη. Η στρατηγική της μπορεί να ε, βοηθήσει. Όλοι έχουν ως στόχο να μεγεθύνουν την ε, περιφερειακή προοπτική σε συνεργασία και με άλλα μέρη της Ευρώπης, αλλά για ορισμένες περιφέρειες, αλλά και για τις μητροπολιτικές περιοχές και στο παγκόσμιο επίπεδο. ώστε να μεγιστοποιηθεί η εκμετάλλευση του ευρωπαϊκού δυναμικού. Και νομίζω μάλιστα ότι είναι και σωστό να πει κανείς ότι σε άλλες υπήρους όπως ε, στη Ρωσία, όπως στην Ασία, αυτές αναπτύσσουν στρατηγικές για ολόκληρη την περιοχή τους. Και διαρθρώνουν τις ε, περιοχές τους με σφαιρικότερο τρόπο και αυτό θα πρέπει να κάνει και η Ευρώπη. Θα κάνω μερικές καταληκτικές παρατηρήσεις. Εμείς εδώ βρισκόμαστε ε, μπροστά σας για να βοηθήσουμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της πολιτικής και θα χαρούμε πολύ να δούμε εκδήλωση ενδιαφέροντος και από τη δική σας Επιτροπή για πιο συγκεκριμένα θέματα βεβαίως εφόσον αυτά θα είναι Έτοιμα να συμμετάσχετε σε κάποιες από τις εκδηλώσεις που θα ε, οργανώσουμε ώστε να συναθρήσουμε επιστήμονες, πολιτικούς υπευθύνους και ούτω καθεξής για να συνεργαστούν. Θα κάνουμε και δημοσιεύσεις που ίσως σας ενδιαφέρουν. Θα πρέπει να μου δώσετε τις απόψεις σας, το λεγόμενο ε, feedback. Τέλος, η ΕΣΠΟΝ είναι πρόγραμμα των διαρθρωτικών ταμείων. Ταυτόχρονα αποτελεί και ένα είδος παρατηρητηρίου για τις ε, τάσεις και την δυναμική που αναπτύσσεται στις περιφέρειες. Γνωρίζουμε ότι από το πολιτικό επίπεδο κάποιοι είπαν ότι ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει ίσως μια συνέχεια ε, στην προσπάθεια παραγωγής δεδομένων που έχουν σχέση με τις περιφέρειες και τα κέντρα και τα μετροπολιτικά κέντρα κτλ. Αυτό ίσως είναι κάτι το οποίο πρέπει από τώρα να εξεταστεί. Η λογική των διαθωτικών ταμείων που λέει ότι πρέπει να σταματά το πρόγραμμα για δύο χρόνια και μετά να ξαναρχίζει που το είδαμε και όλα τώρα, δεν είναι σωστή λογική. Και πάντως όχι για κάτι το οποίο θα πρέπει να έχει ως στόχο να προσφέρει στο πολιτικό επίπεδο μια διαρκή ροή πληροφοριών, ώστε να μπορούν οι πολιτικές αποφάσεις να λαμβάνονται ε, στην βάση των πληροφοριών αυτών και με ε, τρόπο παραγωγικό. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και βεβαίως η ιστοσελίδα μας είναι πάντα στη διάθεσή σας. Είναι πολύ ε, πλούσια και βεβαίως είναι απολύτως δωρεάν διαθέσιμη σε όποιον ενδιαφέρεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μέλμπι για όσα μας είπατε. Μεταξύ αυτών ορισμένα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και νέα για μένα, δεν τα γνώριζα. Δεν ανέμενα δηλαδή να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο να ασχολείται με τις περιφερειακές επιπτώσεις, δηλαδή τις επιπτώσεις της περιφέρειας της αύξησης των τιμών της ενέργειας, καθώς επίσης για τα δημογραφικά κλπ. Υπάρχουν ορισμένες πληροφορίες οι οποίες ακόμα δεν είναι γνωστές στην Επιτροπή μας και βεβαίως μπορείτε να μας τις διαθέσετε εφόσον τις ζητήσουμε. Πράγματι. Τώρα, ερωτήσεις ή σχόλια των συναδέλφων. Κύριε Βανίστερόι, Λαμπέρ, εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, εντυπωσιάστηκα από την ποσότητα των πληροφοριών, των δεδομένων τα οποία μας δώσατε. Έχω βέβαια και κάποιες ερωτήσεις. Εδώ στο Κοινοβούλιο φτιάχνουμε το πρόγραμμά μας και εμείς έχουμε τη ΣΤΟΑ που ασχολείται με τα επιστημονικά, έχουμε διάφορα τέτοια, διάφορες τέτοιες ομάδες και καλό είναι να υπάρχει κάποιος συντονισμός ανάμεσα στα διάφορα αυτά όργανα για να ξέρουμε τι να βάλουμε εμεί στο πρόγραμμά μα ανάλογα με το τι ήδη υπάρχει. Για παράδειγμα στην ΕΣΠΟΝ, όπω μα είπατε, και να μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τα δικά σα στοιχεία και να τα συμπεριλαμβάνουμε στο δικό μα πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, λέτε ότι δυσκολεύεστε με το θέμα της χρηματοδότησης στην Ευρώπη ανάλογα με την προγραμματική περίοδο. Εσείς έχετε ένα προπολογισμό για να καταλήξετε στα δεδομένα σας. Πιστεύετε λοιπόν ότι με τη συνθήκη της Λισαβόνας αυτή η εδαφική συνοχή που γίνεται πάλι στόχος μπορεί να βοηθήσει περισσότερο. Και πιστεύετε ότι πρέπει ο στόχος αυτός να γίνει πιο συγκεκριμένος. Μας δείξατε ένα σωρό χάρτες που ερμηνεύουν την κατάσταση μέσα στην Ευρώπη. Είναι καλό γιατί βλέπουμε έτσι σε περιφερειακό επίπεδο τι πάει καλά τι πάει λιγότερο καλά, τι δυνατότητες υπάρχουν. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να συνδυάσουμε τα στοιχεία που έχουμε με τους χάρτες αυτούς που μας παρουσιάσατε για να οργανώνουμε και εμείς τις εργασίες μας. Τώρα συγκεκριμένη ερώτηση. Τέλος. Όσον αφορά την ατζέντα της Λισαβόνας και τις επενδύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα για την έρευνα. Θεμελιώδης έρευνα, εφαρμοσμένη έρευνα. Σε περιφερειακό επίπεδο τι ισχύει, γιατί δεν είδα να μας λέτε κάτι γι' αυτό πολύ. Θα ήθελα να ξέρω σε περιφερειακό επίπεδο τι γίνεται με την έρευνα και την ανάπτυξη και γενικότερα με την ατζέντα της Λισαβόνας. Πάντως εκτιμώ ιδιαίτερα τη δουλειά σας και θα ήθελα να σας ξαναδώ, γιατί μας βοηθάτε στο έργο μας. Ευχαριστώ. Μπορείτε να απαντήσετε αμέσω. Έχουμε κάποιο χρόνο στη διάθεσή μα, ώστε ε, μπορείτε να απαντάτε και απευθεία. Ναι, θα προσπαθήσω. Χαίρομαι πρώτα απ' όλα που αυτά που σας παρουσιάζουμε σας ενδιαφέρουν και ότι πιστεύετε ότι είναι σημαντικά. Και εμείς πιστεύουμε ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην ολοκληρωμένη προσέγγιση που έχουμε ε, παρατηρώντας τις εξελίξεις, δημιουργώντας στρατηγικές για διάφορες περιφέρειες. Το θέμα της ενέργειας σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό για να υπάρχει περιφερειακή ισορροπία στην Ευρώπη. Υπάρχουν ε, ε, μέρη που έχουν από παλιά παραγωγή, μηχανισμούς, υποδομή αλλά κτίρια τα οποία δεν είναι καλά μονομένα. Σίγουρα και οι τιμές αλλάζουν, αλλού είναι πιο ψηλές, αλλού όχι, οπότε περιφερειακά υπάρχει διαφορά. Τώρα συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Φανίστερόη για αυτό που είπε για την εδαφική συνοχή, ότι χρειάζεται συνεργασία και ότι χρειάζεται μια συνεχή παρατήρηση. Χρειάζεται συζήτηση και να κοιτάμε από κοντά πώς θα οργανώνουμε αυτή την ανάλυση. Τα τελευταία χρόνια έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν διαφορετικές πρωτοβουλίες που προσπαθούν να δημιουργήσουν τη γνώση που χρειάζεται η ΕΣΠΟΝ και όσον αφορά προγράμματα έρευνας. Ξέρω ότι και το Κοινοβούλιο έχει κάνει μελέτες χρησιμοποιώντας τους καλύτερους ερευνητές από την ΕΣΠΟ. Επίσης η Γενική Διεύθυνση Ρέγγιο επίσης ε, για να κάνει αναλύσεις και στατιστικές. Ο στόχος λοιπόν της συνοχής αναφίβολα δημιούργησε μεγάλο ενδιαφέρον στον τομέα αυτό της έρευνας. Όπως είπατε πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να καταλαβαίνουμε τι ακριβώς έχουμε, να αποφεύγουμε τις επικαλύψεις, το θέμα των κονδυλίων είναι θέμα δικό σα. Πάντως το τελευταίο που ρωτήσατε είχε να κάνει με την έρευνα και την ανάπτυξη, τις επενδύσεις εκεί. Εμείς ενημερώνουμε τον χάρτη δικτών της Λισαβόνας για να δούμε πώς αναπτύσσονται οι δίκτες αυτές. Από το 2000 μέχρι το 2006 περίπου μπορούμε να το κάνουμε με τα στοιχεία που μπορούμε να έχουμε. και θα μπουν και αυτά τα στοιχεία στην παρατήρηση που γίνεται την Οικοσασέλιδη και θα τα έχουμε τον Απρίλιο της επόμενης χρονιάς. Θα πρόκειται λοιπόν για νέα ενημέρωση και εσείς μπορείτε έτσι να μάθετε ποια είναι η περιφερειακή κατανομή όσον αφορά τις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Το 2007 πάντως ήταν προφανές, συγγνώμη, το 2000 διορθώνω μιλητής, το 2000 ήταν προφανές ότι οι βόρειες περιοχές και εκείνες που βρίσκονται μέσα στο Πεντάγωνο ήταν εκείνες που έδιναν μεγαλύτερες επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Ευχαριστούμε. Κωνσταντ Σκρέλ. Στο παρελθόν και μάλλον με συμπτωματικό τρόπο, τυχαίο τρόπο δηλαδή, είχα συναντήσει εκπροσώπους του ΕΣΠΟΝ και κάθε φορά, όπως και σήμερα, εξεπλάγει από το πλήθος των δεδομένων που μπορεί να προσφέρει το ΕΣΠΟΝ. Και κάθε φορά θεωρούσα ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιητικό να μην τα λαμβάνει τα στοιχεία αυτά η <clears throat> Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, διότι ομολογώ ότι δεν σκέφτομαι να πάσα στιγμή ότι μπορώ να πάω στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΟΝ για να ε, ε, βρω εκεί δεδομένα τα οποία μπορώ να χρησιμοποιήσω για την εργασία μου. Θα ήταν λοιπόν ιδιαίτερα καλό να λαμβάνουμε τακτικά τις δημοσιεύσεις σας και όχι απλώς την υπόμνηση ότι υπάρχει στο σελίδα σας. Και όχι μόνο α, πίνακες αριθμών, αλλά και οπτική εικόνα σε χάρτες που καθιστούν περιττές τις μακρές συζητήσεις. Και επειδή χθε μιλήσαμε για ένα μη έγγραφο το οποίο λάβαμε για τη μελλοντική διαρθρωτική πολιτική, αυτό δείχνει πόσο ενδιαφέροντες είναι οι χάρτες αυτοί που μας δείξατε, διότι αφενός δείχνουν ότι δεν έχει νόημα πραγματικά να κάνουμε συγκέντρωση της ε, πολιτικής συνοχής σε 10 χώρες μέλη, αλλά ότι πρέπει να δούμε την Ευρώπη ως αυτό που είναι, δηλαδή πολύ πιο ποικίλη και διαφορετική. Και γι' αυτό θα χαρώ ιδιαίτερα εάν έχουμε περισσότερες πληροφορίες εκ μέρους σας και περισσότερες δημοσίευσεις. Έχω μια απλή, ίσως λίγο ανόητη ερώτηση προς το τέλος. Σε κάθε χάρτη σας λέτε ότι ο χάρτης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι απηχεί την άποψη της Monitoring Committee έχετε πάντοτε σε ένα κουτάκι εκεί από κάτω αυτή την φράση. Αυτό τι σημαίνει, ότι υπάρχει δυνατότητα διαφορετικής ερμηνείας των αριθμών όπως θέλει ο καθένας ή σημαίνει ότι ναι μεν οι αριθμοί είναι αυτοί αλλά πολιτικά θα θέλαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μόνο οι βουλευτές είναι υπεύθυνοι για τα όσα λένε. Οι επιστήμονες μπορούν πάντοτε να κρυφτούν πίσω από τα δεδομένα. Αυτό ως ε, σχόλιο. Αλλά κοιτάξτε, έχουμε τόσα πολλά θέματα από την αλλαγή του κλίματος μέχρι την ασφάλεια της προμηθείας της ενέργειας, μέχρι την προστασία των εδαφών κλπ. που έχουν σχέση και με τα περιφερειακά. Που μάθαμε σήμερα ότι υπάρχει μια ε, πηγή ε, πληροφοριών και δεδομένων και πράγματι δεν υπάρχει αυτοματισμός για το πώς θα διαθέτουμε τα ε, δεδομένα αυτά, θα πρέπει εμείς να τα αναζητούμε. Πράγματι, όμως αν είχαμε ε, κάπως αυτόματη διάθεση το ε, διαβίβαση των δεδομένων αυτών, αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ. Παρακαλώ κύριε Μελμπή, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για τα θετικά σας λόγια. Όσον αφορά την ενημέρωσή σας και της Επιτροπής σας είναι κάτι που μπορεί πάρα πολύ εύκολα να τακτοποιηθεί στην πράξη. Εάν θέλετε, εμείς μπορούμε να φροντίσουμε να παίρνετε πάντα ε, αρκετέ εφαρμογές κάθε φορά που έχουμε δηλαδή ένα νέο θέμα να ενημερωνόσαστε, να το παίρνετε, να σας το μοιράζουμε και να σας δίνουμε τουλάχιστον ε, μερικά από τα νέα αντίγραφα, δύο αντίγραφα τουλάχιστον να σας δίνουμε για να μπορείτε να κοιτάζετε και τις εκθέσεις σύνθεσης που ήδη υπάρχουν και ό,τι καινούριο έρχεται. Έχουμε και κάποιο newsletter το οποίο ίσως μπορούμε να το στέλνουμε στη γραμματεία σας προς ενημέρωση. Έτσι ενημερώνεστε για το τι συμβαίνει, τι φτιάχνουμε, με τι ασχολούμαστε κάθε φορά. Τώρα όταν μιλάτε για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Ε, βέβαια, αυτό είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα, διότι όλοι γνωρίζουν ότι πάντα υπάρχει μια δυνατότητα, αν θέλει κανείς για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, τα στοιχεία μπορεί πάντα να αλλάξει χάρτες, ταξινόμηση, μπορεί πάντα να συνδυάσει δείκτες στους χάρτες κλπ. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα έτσι, μαγειρέματος των αποτελεσμάτων αν θέλετε. Όμως εδώ είμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε μια ηθική προσέγγιση. Προσπαθούμε δηλαδή να δίνουμε την πληροφορία που η πεποίθησή μας είναι ότι παρουσιάζεται με τον καλύτερο τρόπο. Πάντα υπάρχουν δυνατότητες κανείς να ερμηνεύσει τα πράγματα και να επικρίνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ένα χάρτη. Αυτό είναι σίγουρο. Σε διάφορους βαθμούς μπορεί να αλλάξει την κλίμακα για παράδειγμα σε ένα χάρτη και άλλα πράγματα μπορεί να κάνει κάτι το οποίο αλλάζει τελικά την εικόνα. Αλλά πρέπει να πιστέψετε ότι εμείς χρησιμοποιούμε τους καλύτερους επιστήμονες στην Ευρώπη και προσπαθούμε να κρατήσουμε και υψηλότατο επίπεδο επιστημονικής ηθικής. Προσπαθούμε να παρουσιάζουμε τα πράγματα με σοβαρό τρόπο. Ευχαριστούμε. Τώρα, στο κύριο Σκύριλοφ να έχει χρόνο για την έκθεσή θα δώσω το λόγο στον κύριο Κόρτες για την ερώτησή του. Μετά στον κύριο Πλάσετ και Αλφουσί. Λοιπόν, ναι, Πρόεδρε, συγγνώμη, συγγνώμη, ακούγεται από την αίθουσα. Μάλλον με λάθος σειρά ξεκίνησαν ομιλητές. Πρώτα ο κύριος Κορτές, λέει ο Πρόεδρος. Πρώτον, σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά σας. Είναι πολύ σοβαρή δουλειά, πραγματικά. Δουλειά που μας ε, διευκολύνει, μας παρουσιάζει έτσι μια αντικειμενική εικόνα της Ευρώπης στην οποία βρισκόμαστε. Μας βοηθάει επίσης την Επιτροπή μας να καταλάβει καλύτερα, να αναλύσει καλύτερα και να πάρει καλύτερες αποφάσεις στο μέλλον. Διαπιστώνω ότι υπογραμμίζεται πολιτικές ε, για το μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, την αύξηση του πληθυσμού, ενέργεια, πράγματα καυτά για το μέλλον της Ευρώπης είναι όντω πολιτικές του μέλλοντος. Αυτό όμω που διαπιστώνω, για να πω και κάτι, είναι χάρτες που έγιναν το 2000 δεν θα έπρεπε να υπάρχει ενημέρωση της τεκμηρίωσης αυτής. Δεν θα έπρεπε να είναι όσο γίνεται πιο κοντά στη σημερινή ημερομηνία. Καταλαβαίνω ότι η δουλειά είναι σύνθετη και δύσκολη, αλλά καλό θα ήταν η Επιτροπή μας να έχει όσο γίνεται πιο ενημερωμένα στοιχεία. Σημερινά ή δυνατόν. Και να ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο γιατί δεν το είδα στα έγγραφά σα. Πρόκειται για την απασχόληση ή καλύτερα την ανεργία. Υπάρχουν στην ΕΣΠΟΝ στοιχεία όσον αφορά την ανεργία, την απασχόληση ενημερωμένα και αν υπάρχουν, εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να τα έχω. Και κάτι ακόμα να ρωτήσω. Πώς βλέπετε εσείς τους δείκτες που χρησιμοποιείτε για να μετρήσετε την ε, προσβασιμότητα με τρένο ή στις ενέργειες μεταφορές. Εσείς αυτούς τους δείκτες πώς τους βλέπετε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βλάσακ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση αυτή και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ σε ένα πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε δει πολλούς χάρτες, πολλά σχέδια με στοιχεία δεδομένα από το 2000-2005. Για μας την Επιτροπή αυτό είναι ζωτική σημασίας να έχουμε όσο γίνεται πιο ενημερωμένα στοιχεία, δηλαδή το 2006-2007 καλύτερα. Γιατί έτσι μόνο μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά μέσα στην ε, δομή που έχουμε. Επίσης, το ζήτημα είναι κατά πόσο θα ήταν δυνατόν στους χάρτες αυτούς να συμπεριλάβουμε και τους κατάλληλους δείκτες που μας βοηθάνε να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει ο χάρτης. Εσείς μας μιλήσατε και για το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε. Θέλουμε επίσης να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα, ε, την απόδοση των κονδυλίων που πηγαίνουν σε αυτό το στόχο. Όπως επίσης και για την ενέργεια. Θέλω να ξέρω κατά πόσο εσείς έχετε πληροφορίες για την μέτρηση της εξοικονόμησης ενέργειας. η εφαρμογή νέων μέσων μόνωσης κτηρίων κλπ. And Mr. Alfuzi, Κύριε κύριος τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Όντω και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ το έργο σας. Εννοείται, η Επιτροπή μας ενδιαφέρεται γι' αυτά. Το πρώτο τώρα που θέλω να πω είναι οι χάρτες που μας παρουσιάσατε έχουν και πολιτικό νόημα, όχι μόνο τεχνικό, γιατί μας επιτρέπουν να καταδείξουμε τις προθέσεις της Επιτροπής που ανακαλύψαμε χθε όσον αφορά την πολιτική συνοχής δείχνουν ποια είναι η κατάσταση σε περιφερειακό επίπεδο και δείχνουν ότι πρέπει να υπάρχει μια περιφερειακή διάσταση στην πολιτική συνοχή. Ελπίζω να του δει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκείνοι που εκπονούν την μελλοντική πολιτική συνοχή. Επίση, το έργο σα μα βοηθάει να προσεγγίσουμε και να διευκρινίσουμε περισσότερο τη δουλειά που εμεί θέλουμε να κάνουμε για την εξέλιξη των δικτών. Βλέπετε ότι εμεί έχουμε πάντα το δίκτυο του Εδάφου και του ΑΕΠ είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτούς. Εσείς με τις εργασίες σας έχετε βρει δείκτες οι οποίοι θα μπορούσαν να ήταν ενδιαφέροντες για μας, προκειμένου να μπορούμε έτσι καλύτερα να αντιληφθούμε πώς προχωράει η περιφερειακή εξέλιξη πέρα από το ΕΠ. Και κάτι άλλο που μας απασχολεί είναι οι διαφορές που υπάρχουν μέσα στον ίδιο χώρο. Μερικές περιφέρειες είναι κατακαιρματισμένες. Για παράδειγμα, όταν περνάμε από το Παρίσι, μια αστική περιοχή με αριστεία πανεπιστημίων κτλ. και πάμε λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα, διαπιστώνουμε ότι η κατάσταση είναι διαφορετική. Και αυτές οι διαφορές που εντοπίζονται είναι ανησυχητικές. Και δεν είναι μόνο στον αστικό χώρο, αλλά και στην Ήπεθρο. Υπάρχουν ε, χώρες, στην, ε, μάλλον, συγγνώμη, περιφέρειες στην Ήπεθρο, όπου κάπου υπάρχει ανάπτυξη στη Γεωργία, κάπου αλλού αντίθετα εγκαταλείπει ο κόσμος. Είναι κατακαιρματισμένες δηλαδή, δεν είναι ενιαία μια περιφέρεια, δεν είναι ομοιόμορφη. Ευχαριστώ. Κύριε Μέρμπη, θα θέλατε να απαντήσετε και σας παρακαλώ να είσαστε σύντομος γιατί περνάει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Ευχαριστώ. Προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομο, απαντώντα πολύ καλέ ερωτήσει. Βέβαια, η απασχόληση και η ανεργία αποτελούν στοιχεία και δείκτες που παρακολουθούμε. Είναι απλές αυτές οι πληροφορίε. Ίσως μπορούμε να το συνδυάσουμε με το γεγονό ότι χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν πιο επικαιροποιημένα στοιχεία, διότι έχει πρόβλημα η Ευρώπη. Έχουμε πρόβλημα διότι δεν έχουμε περιφερειακά στοιχεία που να καλύπτουν όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Εδώ ίσως ε, μπορούμε να κάνουμε κάτι, ίσως να ε, λάβει τη μορφή αιτήματο αυτό. Ε, θέλουμε περιφερειοποιημένες πληροφορίες για το 2006-2007 και ίσως και αργότερα, αλλά είναι αδύνατο να βρούμε τα στοιχεία. Δεν μας τα δίδει η Eurostat γρήγορα, διότι είναι μακρά η διαδικασία ε, στάθμισης των στοιχείων ε, και επεξεργασίας τους. Εξετάζουμε περιβαλλοντικά θέματα. Δεν νομίζω ότι έχει αποφασιστεί ακόμα από πλευράς Επιτροπής Ελέγχου να προβεί σε έρευνα σχετικά με το πώς τα επενδυθέντα ποσά δημιούργησαν θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και για εξοικονόμηση ενέργειας. Ίσως αυτό να αφορά περισσότερο τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο να προβεί σε αυτού του είδους την ανάλυση όσον αφορά τις διάφορες ε, παρεμβάσεις. Εγώ θα έλεγα ότι όσον αφορά τους δείκτες, οι δείκτες όσον αφορά την πρόσβαση είναι δείκτες που προσπαθούν από κάθε σημείο, κάθε περιοχή, κάθε περιφέρεια στην Ευρώπη, από σημεία περιφερειών στην Ευρώπη, να δουν πόσος χρόνος απαιτείται για να πλησιάσεις συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων. Και έτσι οδηγούμαστε στους χάρτες που βλέπετε στην οθόνη. Η προσβασιμότητα μπορεί να μετρηθεί ποικιλοτρόπως. Αυτό είναι σίγουρο. Θεωρήσαμε όμως ότι είναι ένας καλός τρόπος αυτός, ασφαλής τρόπος για να δίνουμε πληροφορίες για τον τόπο και την προσβασιμότητα. Αλλά πρέπει να δούμε ότι οι χάρτες κάνουν προσμέτρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένα σημείο από κάθε περιφέρεια δίνει τιμή, η οποία τιμή εισάγεται στο χάρτη. Όσον αφορά το ΑΕΠ, θα ήθελα να πω ότι όλοι συμφωνούν σήμερα ότι χρειάζεται οριζόντια προσέγγιση όσον αφορά την ανάπτυξη των περιφερειών. Δηλαδή, χρειάζεται ποικιλία πληροφοριών, μεγάλη, μεγάλη ποικιλία δικτών, οι οποίοι δείχνουν πολλά ισχυρά και αδύνατα σημεία περιφερειών. Γίνεται σύγκριση μεταξύ περιφερειών της Ευρώπης βάσει δικών μας πληροφοριών και άλλων πληροφοριών. Και το ΕΠ ίσως τώρα έχει την καλύτερη χρήση όσον αφορά την διανομή των πόρων. Αλλά όταν πρέπει να δαπανηθούν οι πόροι χρειάζεται πολύ ευρύτερη προσέγγιση και ελπίζω το μήνυμα να είναι ξεκάθαρο όσον αφορά το τελευταίο στοιχείο, όσον αφορά το διαχωρισμό μεταξύ περιφερειών που είναι τα όρια. Δεν είμαστε πολύ καλοί σε αυτό, διότι αυτό το αφήνουμε σε εθνικές και περιφερειακές δραστηριότητε και αναλύσεις. Αποστολή μας είναι να δούμε το ευρωπαϊκό, την ευρωπαϊκή εικόνα, να δούμε τι δυναμική υπάρχει, ποιες τάσεις υπάρχουν ποιες προοπτικές υπάρχουν για όλη την Ευρώπη. Οπότε αυτό μας οδηγεί σε όρια όσον αφορά τις περιοχές στις οποίες μπαίνουμε. Η στοχευμένη ανάλυση που αναφέραμε και η δυνατότητα να μπαίνουμε σε λεπτομέρειες, σε διάφορες συγκεκριμένες μελέτες, αυτό έχει αναλυθεί σε διάφορα προγράμματα, αλλά δεν είναι ο δικός μας βασικός στόχος να μπούμε σε λεπτομέρειες όσον αφορά τις περιφέρειες. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Σακέντη ας υποβάλει το ερώτημά του. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να απευθύνω σε ευχαριστίες μου για τη ρεαλιστική προσέγγιση που παρουσιάστηκε στην παρουσίαση που έγινε. Καμιά φορά αντιμετωπίζουμε δεδομένα τα οποία μας συγκλονίζουν και δεν τα γνωρίζαμε. Το κόμμα μου, το Γιόμπικ, είναι ε, μια ευρωσκεπτικιστική ε, πολιτική δύναμη. Δεν το κρύβουμε, αλλά σαν ευρωβουλευτής εκπρόσωπος του κόμματος φοβούμε ότι η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της μόνο ενωμένη, με έναν ενίο τρόπο. Τα προβλήματα δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν όμως από τις Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης, από μια Ευρώπη όμως των εθνών. Και αυτή η Ευρώπη των κρατών ε, χρειάζεται έναν ισχυρό ευρωπαϊκό συντονισμό. Τις πρόσφατες εβδομάδες επισκέφθηκα ουγγρικές περιφέρειες και την Τανσιλβανία και τη Ρουμανία επισκέφθηκα και εκεί εξέτασα διάφορα προγράμματα που υλοποιούνται. Και βρήκα, διαπίστωσα ότι υπάρχει έλλειψη ευαισθητοποίησης όσον αφορά τους μελλοντικού κινδύνους που ίσως ελοχεύουν. Και οι ντόπιοι δεν είναι έτοιμοι για αυτούς τους κινδύνους. Μπορεί για να είναι προφανής η κίνδυνη, αλλά στην Ανατολική Ευρώπη και στα νέα κράτη-μέλη δεν είναι καθόλου έτοιμοι οι άνθρωποι για μελλοντικέ απειλές δεν υπάρχει εμπειρία, δεν υπάρχουν οι ρουτίνες που έχουν δημιουργήσει τα παλιά κράτη-μέλη. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα ήταν σημαντικό να υπάρχει μια θέση της Επιτροπής μας, μια στάση της Επιτροπής μας όσον αφορά τις περιφέρειες της Κεντρικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Έχω επίσης και ένα ερώτημα. Ο μιλητής αναφέρθηκε στο ότι η Ευρώπη ίσως να ε, αντιμετωπίσει εθνοτικές συγκρούσεις λόγω μεταναστεύσεων και κυρίως στις νότιες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχετε κάνει κάποιους υπολογισμούς όσον αφορά τις περιφέρειες κυρίως της νότιας Ευρώπης που αλλάζουν οι εθνοτικές ισορροπίες στο μέλλον. Η μετανάστευση φαίνεται ότι ίσως να αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που ίσως να αλλάξει τις εθνοτικές ισορροπίες σε κάποιες περιοχές. Καλώς, ευχαριστώ. Ο κύριος, ο κύριος Ολζενίζακ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Το όνομά μου είναι Όλεν Τσακ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν κύριε Πρόεδρε, αναφέρθηκε η εξειδίκευση των στοιχείων. Στοιχείων ε, που εξετάσατε εσείς. Και είναι ενδιαφέρον να βλέπει κανείς ποιες τάσεις υπάρχουν και ποιες μελλοντικέ προπτικές διαμορφώνονται. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Όταν βλέπει κανείς τα πορίσματα αυτών των ερευνών, και εδώ συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα υπόθηκαν, και όλοι στις συνεδριάσεις και στι συναντήσει που έχουμε στην Ευρώπη βλέπουμε ποια προβλήματα υπάρχουν. Λοιπόν, ξέρουμε ότι είναι πολύ διαφοροποιημένη η Ευρώπη. Υπάρχει ποικιλία. Και όταν μιλάμε για πολιτική συνοχή, εκεί υπάρχουν πολλά επίπεδα. Λοιπόν, το ερώτημά μου που σα έλεγα είναι το εξή. Όταν προσπαθείτε να κάνετε προβλέψει βάσει των υφισταμένων πληροφοριών, μπορείτε να καταλήξετε σε ε, συμπεράσματα λογικά όσον αφορά την παρούσα κατάσταση και μπορείτε να κάνετε διορθώσεις. Νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή... Δεν κάνουν ε, λάθος. Αν έχουν γίνει σφάλματα κατά το παρελθόν, τα σφάλματα πρέπει να διορθώνονται βέβαια. Μπορείτε να μας πείτε, κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα ενδεχόμενα λάθη και εσείς μπορείτε να επηρεάσετε ώστε τέτοια σφάλματα να μην ξαναγίνουν στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Βέλμπη, παρακαλώ να συνοψίσετε την απάντησή σας σε πέντε λεπτά παρακαλώ. Εντάξει. Εγώ δεν μίλησα για εθνικές ε, συγκρούσεις. Εγώ έδειξα απλώς ένα χάρτη που δείχνει ότι ίσως ε, η μετανάστευση στο μέλλον να ενταθεί από τον Νότο. Θα λέγω ότι αυτό είναι το κύριο συμπέρασμά μου από το συγκεκριμένο χάρτη που σας έδειξα. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα για την κατανομή των εθνικών ομάδων στα διάφορα σημεία της Ευρώπης επί του παρόντος. Δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο μέχρι τώρα. Όσον αφορά όμως το θέμα των προβλέψεων, ιστορικών δεδομένων κτλ. Καταλαβαίνω ότι λέτε ότι καλό θα ήταν να έχουμε μια τέτοια διάσταση, μια τέτοια άποψη για το μέλλον. Και εγώ θα έλεγα ότι η ΕΣΠΟΝ μέχρι τώρα έχει χρησιμοποιήσει ένα σενάριο που υποθέτω ότι θα μπορούσε να είναι πολύ ενδιαφέρον ε, και για να έχετε εσείς περισσότερες πληροφορίες για το πώς δουλεύουμε. Είναι ένας αρκετά κλασικός τρόπος. Παίρνουμε ε, μια μεθοδολογία στρατηγικού σχεδιασμού, αξιολογούμε την κατάσταση, είτε ιστορικά μπορεί κανείς να το δει, ποιες είναι οι τάσεις δηλαδή που είχαμε τα τελευταία 10 χρόνια, και έτσι μπορείτε να κάνετε μια πρόβλεψη βάσει αυτών των ιστορικών δεδομένων. Δημογραφικά στοιχεία κλπ. Αλλά μετά πρέπει να προσπαθήσετε να προκαταλάβετε την κατάσταση για το μέλλον. δείτε δηλαδή ποιε άλλε δυνάμει λειτουργούν, ποιε άλλε παράμετροι παίζουν ρόλο για τη διαμόρφωση της κατάσταση στο μέλλον. Και αυτό σα έδειξε και από την αρχή με τι διαφάνειε. Βάσει αυτού λοιπόν μπορείτε να καταλήξετε και σε αντιφατικά σενάρια που μπορεί να δείχνουν πιο ανταγωνιστικό προσανατολισμό ή μεγαλύτερη συνοχή. Τα δύο άκρα. Οπότε διαφοροποιείται πολύ κατάσταση. Γιατί όταν υπάρχει μεγάλη ανταγωνιστικότητα μπορεί να υπάρχει μεγάλο ΕΠ. Αλλά θα περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή μέσα στην Ευρώπη, σε κάποια καυτά σημεία. Ενώ όταν καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι έχουμε περισσότερο πολιτική συνοχής, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει καλύτερη κατανομή. Αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο ίσως ΑΕΠ. Αυτό, θέλετε, ήταν και ένα από τα κύρια βρήματά μας. Εγώ ευχαρίστω σας δίνω το έγγραφο, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι από τη στιγμή που έγινε, μετά είχαμε την οικονομική κρίση, η οποία προφανώς και δημιουργεί μια νέα κινητήρια δύναμη, που αλλάζει κάπως το σενάριο. Άρα χρειάζεται κάποια αναθεώρηση του σενάριου μας, γιατί πρόκειται για μια εξέλιξη που βέβαια είχε μεγάλο αντίκτυπο στην κατάσταση. Ωραία, για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας, για τα όσα μας είπατε. Ευχαριστούμε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Ερχόμαστε και πάλι στο σημείο 7. Πάμε πίσω δηλαδή. Και θέλω να δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ευγένη Κύριλοφ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δυστυχώς δεν έχω και πολλά να σας πω, δηλαδή δεν έχουμε τίποτα φοβερές εξελίξεις. Από την προηγούμενη συνεδρία της Ρέζιο είχαμε δύο συναντήσεις στο Συμβούλιο στις 8 και στις 27 Οκτωβρίου αντίστοιχα, όπου συζητήθηκαν οι τροπολογίες του Γενικού Κανονισμού για τα Ερθωτικά Ταμεία. Επετεύχθη κάποια πρόοδος μετά την παρουσίαση ενός non-paper από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ γι' αυτό την Επιτροπή. Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει ακόμα κοινή θέση από πλευράς του Συμβουλίου. Το non-paper θέλει να προσθεθούν δύο στοιχεία. Αντικαθίσταται η αρχική πρόταση όσον αφορά το άρθρο 7, ε, 77 που έχει να κάνει με τη συγχρηματοδότηση. Έπειτα υπάρχει το θέμα της ρευστότητα που προσπαθεί και αυτό να το καλύψει μέσω του κοινωνικού ταμείου με 2% του περιφερειακού ταμείου. Συν βέβαια την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Έπειτα υπάρχει τροποποίηση του 82. Και η δεύτερη αλλαγή έχει να κάνει με την αναβολή κατά ένα χρόνο της υποχρέωσης του αυτόματου κανόνα. Όσον αφορά την Επιτροπή, έτσι, τα προγράμματα τα οποία εγκρίνονται το 2007 έχουν ένα χρόνο παραπάνω στη διάθεσή τους για να προχωρήσουν σε εφαρμογή διατηρώντας την δημοσιονομική πειθαρχία. Νομίζω ότι αυτή η ελαστικότητα είναι αναγκαία, δεδομένου ότι έτσι, όπως ξέρουμε, μπορεί να ξεκινήσει το πρόγραμμα και να συνεχιστεί και μετά το 2007. Βέβαια αυτό απαιτεί το τροποποίηση του άθρου 93. Οι πρόσφατες συζητήσεις στο Συμβούλιο πλησίασαν συμφωνία όσον αφορά ε, την απλούστευση που απαιτείται και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται. Το πιο δύσκολο είναι οι προκαταβολές και ίσως αυτό το στοιχείο να εγκαταληφθεί ούτω ώστε να επιτευχθεί συμφωνία επί των υπολείπων. Η επόμενη συνεδρίαση του Συμβουλίου σύντομα θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου και αν υπάρξει θετικό αποτέλεσμα στην Ολομέλεια την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου μπορούμε να εξετάσουμε ε, το ενδεχόμενο ενό σχεδίου κειμένου της Επιτροπής μας στις συνεδρίες του Δεκεμβρίου. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ανησυχώ, πρέπει να σας το πω αυτό, διότι αυτή η καθυστέρηση εν μέσω της κρίσης που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες δεν είναι κάτι ευπρόσδεκτο καθόλου και θα πρέπει να εκφράσουμε κάποιες ανησυχίες στο Συμβούλιο. Διότι όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, αν αυτό γίνει σε μερικούς μήνες, αν αργήσουν τα μέτρα δεν θα έχουν τα ευταία αποτελέσματα για την αντιμετώπιση της κρίσης. So, Αυτές είναι οι πληροφορίες που ήθελα να σας δώσω και στο Συμβούλιο θα παρακολουθήσω τις ε, επικείμενες διαπραγματεύσεις του σύνεγγης. Okay. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ κύριε Κυρίλοφ. Ας συζητήσουμε σύντομα λοιπόν το θέμα παρακαλώ. Πολύ σύντομα θα ήθελα να πω ότι έχουμε, έχουν αποτελματωθεί οι προσπάθειες, λυπηρό αυτό, διότι περνάμε πράγματι κρίση και θα έπρεπε να μπορούμε να δράσουμε, να κινηθούμε, να αντιδράσουμε εναντί κρίση Χρειαζόμαστε απλούστευση των διαδικασιών, ούτω ώστε να εφαρμοστούν αποτελεσματικά συγκεκριμένα οι παρεμβάσει των διεθνωτικών ταμείων στι επικράτειέ μα. Και θα ήταν σημαντικό να προχωρηθεί το θέμα τώρα. Δεν έχω τίποτα να προχωρήσω. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι, για τη δουλειά που κάνατε. Τη δουλειά που γίνεται από κοινού, μάλλον. Καλώ, ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Η κυρία Σρέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Εκπλήσωμε. Εκπλήσωμε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το θέμα. Κανονικά, για έναν γενικό κανονισμό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταλήγει σε μια αρχική θέση. Και ο εισηγητής την συμπεριλαμβάνει στις διαπραγματεύσεις, ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα να συνδέσει το δικαίωμα ψηφοφορίας του με κάποια από τα κριτήρια. Αυτό δεν συνέβη. Έγινε μια πρώτη συζήτηση και μόνο. Και το ερώτημά μου προς τον εισηγητή είναι το εξής. Ποια σημεία της συζητήσεως μπήκαν στις διαπραγματεύσεις μέσω του εισηγητού. Ήταν δύσκολα τα πράγματα, δεν υπήρχε κάποια θέση της Επιτροπής που συνήθως υπάρχει και νομίζω ότι εμπρότης χρειαζόμαστε ψηφοφορία στην Επιτροπή και μετά να μπορεί να πάει με αυτή τη θέση πίσω του ο εισηγητή τη διαπραγματεύση. Και είναι σημαντικό πριν την προθεσμία του Δεκεμβρίου να έχουμε καταλήξει εμεί σε κάποια θέση. Ε, και είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα, διότι εάν το Κοινοβούλιο πλεί απλώ ότι αποδέχεται τα όσα κάνει το Συμβούλιο και δεν έχει δική του θέση επί κάποιων σημείων το Κοινοβούλιο, είναι δύσκολα τα πράγματα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, α πούμε, απλώς να υπερψηφίσει την επέκταση του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας. Και μόνο. Ε, είναι σημαντικό να διαδραματίσουμε το δικό μας ρόλο στη διαπραγματεύσεις, κάτι που δεν συνέβη μέχρι τώρα. Δεν μπορούμε να έχουμε τον εισηγητή μας να επομίζεται τα πάντα και να προχωρά χωρίς να έχει πίσω του μια θέση του Κοινοβουλίου και άποψη του Κοινοβουλίου που θα πρέπει να συμπεριληφθεί στις συζητήσεις. Υπάρχουν διάφορα θέματα, διάφορα πράγματα που προτείναμε, τα οποία όμως δεν σχολιάστηκαν επουδενή. Πρόεδρος, στην επόμενη συνεδρίαση θα μπούμε σε αναλυτική συζήτηση να δώσω το λόγο στον κύριο Κυρίλοφ για να προβεί σε κάποια σύντομα σχόλια. Ευχαριστώ Πρόεδρε πολύ σύντομα να απαντήσω στην κυρία Σρέντερ. Ξέρετε βεβαίως ότι δεν είμαστε ακόμα εντός της συνθήκης της Αβώνας αν καθυστερήσουμε αν αργήσει η όλη ιστορία μπορούμε να παίξουμε το ρόλο μας που απορρέει από τη συνθήκη. Ε, τώρα πρέπει να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη. Το συζητήσαμε, παρακολουθήσαμε τις εξελίξεις αλλά όπως είπατε είναι θέμα τοποθέτηση Επιτροπής. Λίγο πολύ ξέρω ποια είναι η θέση των συναδέλφων των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Δηλαδή να υποστηρίξουμε ενεργά τη διαδικασία πλούστευσης. Επανειλημμένα το συζητήσαμε στην Επιτροπή και στην ε, πρώτερη θητεία. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα τις επόμενες μέρες, έχουμε κάθε δικαίωμα να μπούμε σε ενδελεχή συζήτηση και βεβαίως να ξεκινήσουμε να διαδραματίζουμε τον πραγματικό μας ρόλο στην όλη διαδικασία. Καλώς, σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ορίστε, για το τελευταίο ερώτημα. Για ακόμη μια φορά θέλω να πω κάτι. Γνωρίζω και εγώ τη διαδικασία. Κατά το παρελθόν είχαμε κάνει την όλη, το όλο εγχείρημα πολλές φορές. Η διαδικασία είναι η οθετή επιτροπή ψήφισμα που καθορίζει την κοινή θέση και μέσω του ψηφίσματος που εγκρίνεται από την Επιτροπή πριν πάμε στην Ολομέλεια, ο εισηγητής πάει και χρησιμοποιεί αυτή τη θέση. Και αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνέβη τώρα. Τουλάχιστον διεξήχθη συζήτηση. Και κατά τη διάρκεια της συζητήσεως κάναμε κάποιες προτάσεις. Προτείναμε κάποια σημεία τα οποία θα συμπεριλαμβανόταν στο περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων. Και αυτό δεν αντικαπτοτρίζεται καθόλου σε αυτά που άκουσα, σε αυτά που μας είπατε. Βεβαίως, είμαστε 100% υπέρ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, όμως είπαμε, η πλειοψηφία είπε ότι θα πρέπει να ε, πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Βεβαίω αναφερθήκαμε σε διάφορα ζητήματα τα οποία μπορούν να τεθούν στα πλαίσια τη καταπολεμήσεω τη κρίση. Και δεν τα αναφέρατε αυτά. Σε έναν κανονισμό κανονικά είχαμε ψήφισμα που εμπεριείχε διάφορα σημεία, ο εισηγητής έπαιρνε αυτά τα σημεία και πήγαινε στη διαπραγματεύση. Αυτό γινόταν παλιά. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, κάτι αντίστροφα. Αυτό γίνεται όταν ο εισηγητής ξεκινάει τις διαπραγματεύσεις. Το μόνο που μπορώ να κάνω τώρα είναι να προτείνω, να συστήσω, να καταλήξουμε σε ένα ψήφισμα το ταχύτερο δυνατόν το οποίο να περιγράφει τις διάφορες θέσεις του Κοινοβουλίου, το ψήφισμα αυτό, και ο εισηγητής να προχωρήσει μετά στις διαπραγματεύσεις βάσει αυτών των σημείων. Διότι είναι σημαντικό η ψηφοφορία να εξαρτάται από αυτά τα σημεία. Και αυτή είναι η μόνη δυνατότητα που υπάρχει να συμπεριλάβουμε τη θέση μας στις διαπραγματεύσεις βάσει της συνθήκη τη Πρόεδρος, πριν συζητήσουμε λεπτομερώς το θέμα, μπορούμε να το κλείσουμε εδώ και να το συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρίαση εκτενώς. Πάμε στο σημείο 11. Εξωτερική μελέτη για την ανάκτηση των δαπανών των ε, Ταμείων Συνοχής στο κάτι μέλη οικονομική απόδοση των δαπανών στον τομέα της συνοχής στα κράτη-μέλη. Ο κύριος Τζον Μπράντλεϊ από το Δουβλίνο θα μιλήσει πρώτα και ο καθηγητής Γκέρχαρτ Ούντιτ από το Μίνστρο τη Γερμανία και ο καθηγητής Ζάνους Ζαλέσκι από την Πολωνία θα πάρουν το λόγο. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Παρακαλώ λοιπόν για μια σύντομη εισαγωγή, καθηγητά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας. Και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να κάνω εδώ την παρουσίασή μου. Σας παρουσιάζω μια μελέτη την οποία κάναμε μετά από αίτημα του προηγούμενου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ολοκληρώθηκε η μελέτη μας το 2009. Η μελέτη που θα σας παρουσιάσουμε έχει ως τίτλο «Απόδοση, οικονομική απόδοση των δαπανών στον τομέα της συνοχής για τα κράτη-μέλη». Για το πρώτο τμήμα ασχολούμαστε με την τις οικονομικές επιπτώσεις πάνω στη περιφέρεια. Δεν αναφερόμαστε εδώ ιδιαίτερα στους δικαιούχους. Προσπαθούμε να υπογραμμίσουμε την συνεισφορά της πολιτικής συνοχής. Εδώ, κατά πρώτον, θέλουμε να δούμε, όπως είπαμε, τον αντίκτυπο ε, πάνω στους ε, δωρητές, πάνω στους καθαρούς εισφορείς. Είδαμε και πώς επηρεάζει την οικονομική συνοχή, η πολιτική συνοχής. Από ό,τι φαίνεται, πάντως, οι πολιτικές συνοχής εξαιτίας του μεγέθους πρώτα απ' όλα επηρεάζουν τις χώρες δικαιούχους, αλλά εξαιτία των διαφόρων οικονομικών αναλύσεων που γίνονται από την εσωτερική αγορά, υπάρχουν επιπτώσεις και πάνω στους καθαρούς εισφορείς. Μέχρι τώρα δεν είχαμε ποσοτικά αποτελέσματα για το εύρος των επιπτώσεων αυτών, του αντικτύπου αυτού. Χάρη στη μελέτη πάντως που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσπαθούμε να καλύψουμε ένα κενό. Για πρώτη φορά εκφράζουμε ποσοτικά σε ένα πλήρες σύστημα ποιος είναι ο αντίκτυπος πάνω στους καθαρούς εισφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουμε δηλαδή ξεκάθαρα για πρώτη φορά πώς επηρεάζεται η πολιτική πώς επηρεάζεται όλη η οικονομική κατάσταση στις διάφορες χώρες εξαιτίας της πολιτικής συνοχής εξετάζουμε την περίοδο 2000 με 2006. Πριν δηλαδή την διεύρυνση του 2004 είχαμε κυρίως την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Τις ε, χώρες που ήταν πριν στη συνοχή και που ήταν οι δικαιούχοι των χρημάτων της συνοχής. Μετά όμως είχαμε και κάποιες περιφέρειες από την Ιταλία ή τη Γερμανία που επίσης υποφελήθηκαν πολύ από τέτοια κονδύλια. Από το 2004 και μετά βλέπουμε ότι συμπεριλαμβάνονται πια και όλες οι νέες χώρες της πρώτης διεύρυνσης. Η Ρουμανία και η Βουλγαρία όχι ακόμα, δεν λαμβάνονται υπόψη στη μελέτη μας γιατί μπήκαν το 2007 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μελέτη λοιπόν έγινε στα πλαίσια διεθνούς συνεργασίας. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από τον κύριο Μπράντλη, από την Ιρλανδία που ήδη από τη δεκαετία του 80 ασχολείται με τη διαρθρωτική πολιτική. Είναι ερευνητή και μετά είχαμε τον καθηγητή Ζαλέσκι από την Πολωνία. Στην Πολωνία, πριν από την ένταξη της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη είχε ασχοληθεί με την διαρθρωτική πολιτική. Και εγώ Έρχομαι από τη Γερμανία και ασχολούμαι με την γερμανική διαρθρωτική πολιτική ήδη από την αρχή της δεκαετίας του 90. Συνεπώς, η μελέτη που έχουμε εδώ μπροστά μας αποτελεί παράδειγμα διεθνούς συνεργασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δείχνει επίσης πώς μπορούμε μαζί να αξιολογήσουμε την πολιτική συνοχής Μετά από αυτή τη σύντομη εισαγωγή μου θα δώσω το λόγο στον καθηγητή Μπράντλι, ο οποίο θα σα παρουσιάσει την μελέτη και μετά μπορούμε να συζητήσουμε για τα αποτελέσματα τη μελέτη αυτή. Ωραία. Κύριε καθηγητά Ουντίτ, σα ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Μπράντλι τώρα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Τα αποτελέσματα αυτά τα έχουμε ήδη παρουσιάσει το Μάιο στα ευρωβουλευτέ του προηγούμενου κοινοβουλίου. Αλλά μα ζητήθηκε να τα ξαναπαρουσιάσουμε για να τα μάθουν και οι νέοι ευρωβουλευτές. Ελπίζουμε να βρείτε τα αποτελέσματα της μελέτης μας ενδιαφέροντα. Για τους νέους ευρωβουλευτές λοιπόν, ζητάμε Μάλλον για τους παλιούς ευρωβουλευτές ζητάμε κάποια επί και τα έχουν ξανακούσει, αλλά μπορεί να έχουν ερωτήσεις να μας θέσουν. Λοιπόν, μας ζητήθηκε να εκφράσουμε ποσοτικά τις επιπτώσεις της συνοχής, των δαπανών συνοχής, πάνω στους δικαιούχους, στα κράτη δηλαδή, τα οποία επωφελήθηκαν από τα κονδύλια συνοχής, και αυτό για την περίοδο 2000-2006. Μας ζητήθηκε να εκφράσουμε ποσοτικά τα, τις επιπτώσεις επίσης πάνω στους καθαρούς εισφορείς, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεισφορά τους στον ευρωπαϊκό προπολογισμό και πώς επηρεάστηκε το εμπόριό τους. Επίσης μας ζητήθηκε να εντοπίσουμε το μέρος των συμβολέων από τις χώρες δωρητές. Επιτρέψτε μου εδώ να συνοψίσω κάπως τα αποτελέσματα πριν μπω στις λεπτομέρειες. Η ανάλυση μας δείχνει ότι η πολιτική συνοχή εφόσον σχεδιαστεί αποτελεσματικά και εφαρμοστεί σωστά, βοηθάει τον εξυγχρονισμό των χωρών που βρίσκονται πιο πίσω. Δεύτερον, η ζήτηση κατά την περίοδο της εφαρμογής, εδώ η προγραμματική περίοδος είναι 2000-2008, είναι πολύ σημαντική. Όμως η δυνατότητα προσφοράς και τα κέρδη είναι λιγότερα από αυτά τα οποία περιμέναμε. Έπειτα, ο σχεδιασμός της πολιτικής και η εφαρμογή και η απόδοση αυτών δεν είναι τόσο γνωστή. Κάποια τώρα αποτελέσματα αποτελέσματα κλειδί που έχουμε για τις χώρες εισφορής. Ο φόρτος της εισφοράς τους δημιουργεί κάποια μείωση στο ΕΠ και την απασχόληση, πολύ μικρή όμως. Οι χώρες αυτές επωφελούνται από την ε, πολιτική συνοχή στο εμπόριό τους και στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών που βοηθάει την ένταξή τους καλύτερα στην Ευρώπη. Εφόσον εφαρμοστεί και σχεδιαστεί καλά, η συνοχή γενικώ είναι θετική για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερχόμαστε τώρα στο πρώτο ερώτημα. Πόσο μεγάλο άχθος ε, αναλογεί στους καθαρούς εισφορείς. Κάτι ανάμεσα στο 0,1% και το 0,5% του ΑΕΠ των ε, χωρών δωρητών για την περίοδο 2000-2006, κατά μέσο όρο υπάρχει κατανομή. Ο μεγαλύτερος εισφορέας όσον αφορά δηλαδή το μερίδιο στο ΕΠΟ είναι οι κάτω χώρες με 0,5% μετά το Λουξεμβούργο με το 1 τρίτο περίπου, η Γερμανία επίσης και η Σουηδία επίσης. Και ο μικρότερος καθαρός ε, εισφορέας όσον αφορά το ΕΠ είναι η Φιλανδία με 0,1% του ΕΠ. Τι μεγαλύτερε χώρε κάνουν Γερμανία, η Γαλλία, οι κατοχώρε, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που είναι οι μεγαλύτερε χώρε και οι χαμηλότεροι καθαροί εισφορεί είναι, απόλυτοι μάλλον εισφορεί, είναι η Σουηδία, το Βέλγιο, η Ευστρία, η Δανία, το Λουξεμβούργο και η Φιλανδία. Εδώ έχετε ένα πίνακα, ένα διάγραμμα που δείχνει την καθαρή σφορά για ολόκληρη την προγραμματική περίοδο για τη Γερμανία. Βλέπετε την, ε, τις διακυμάνσεις. Όπως επίσης και στη Φιλανδία, όπου το κομμάτι του ΕΠ είναι μικρότερο, γιατί είπαμε ότι είναι από τους μικρότερους καθαρούς ε, εισφορείς. Τώρα, ποιος ε, παίρνει. Και εδώ βάση του ΕΠ. Το μεγαλύτερο μερίδιο κατά αυτή την προγραμματική περίοδο ήταν η Ελλάδα και η Πορτογαλία. Οι πιο σημαντικοί δηλαδή αποδέκτες. Μετά είχαμε Εστονία, Λιθουανία, Λετωνία, Ισπανία, Ουγγαρία, Πολωνία και Μάλτα. Και το χαμηλότερο ποσό Κύπρος, Τσεχία, Σλοβενία, Σλοβακία και Ιρλανδία. Εδώ στο επόμενο διάγραμμα βλέπετε για τις ε, παλιές χώρες, τις πρώτες 15 δηλαδή, ότι η Πορτογαλία παίρνει ένα μεγάλο μερίδιο, περίπου 2% του ΑΕΠ της ετησίως για ολόκληρη την προγραμματική περίοδο και βλέπετε και την Ιρλανδία που ήταν τότε στην διαδικασία απόσυρσης πήρε ένα μικρό κομμάτι. Όσον αφορά τώρα τις 10 χώρες που μπήκαν το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Λετωνία είναι ο μεγαλύτερος δικαιούχος βάσει του ΕΠ και έφτασε 2% τα τελευταία χρόνια της προγραμματικής περίοδου. Είδε Κύπρος που ήδη ήταν μια πλούσια χώρα όταν μπήκε, πήρε ένα πολύ μικρό κομμάτι. Αυτά τα διαγράμματα λοιπόν δείχνουν ότι και από πλευράς ε, άχθους των χωρών δωρητών και από πλευράς κερδών για τους αποδέκτες υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Το επόμενο ερώτημα είναι πώς χρησιμοποιήθηκαν οι δαπάνες της συνοχής. Και εδώ έχουμε χωρίσει το κομμάτι αυτό σε τρία. Τις υποδομές που παίρνουν περίπου το μισό των δαπανών, ανθρώπινοι πόροι που παίρνουν το τρίτο περίπου των συνολικών δαπανών και άμεση αρρωγή στον παραγωγικό τομέα, Γεωργία, 16%. Αν λοιπόν ε, μας ζητάτε να εκφράσουμε ποσοτικά το τι δίνουν οι δωρητές, πρέπει να δούμε πρώτα τι κερδίζουν οι δικαιούχοι, γιατί αυτό είναι το σημείο από το οποίο ξεκινάει η ανάλυση μας. Και πώς το κάνουμε. Υπάρχουν τώρα κάποιες τεχνικές λεπτομέρειε που σας δίνουμε στην έκθεσή μα. Χρησιμοποιούμε οικονομικά μοντέλα έτσι, για να καταλήξουμε στα συμπεράσματά μας. Βλέπουμε πώς λειτουργούν οι χώρε, πώς αντιδρούν στα διευθυντικά ταμεία και γενικότερα στα κονδύλια της συνοχής. Ε, κάνουμε ε, μία εικονική έκφραση για τις δαπάνες αυτές μία προσωμείωση με συνοχή, χωρίς συνοχή και μετά συγκρίνουμε αυτές τις δύο προσωμιώσεις. Και έχουμε και τις δύο προγραμματικές περιόδους, το 2000-2008 και 2009-2020. Η πρώτη δηλαδή είναι η περίοδος εφαρμογής της συνοχής και 2009-2020 χωρίς συνοχή. μετά δηλαδή από την εφαρμογή της πρώτης περίοδου συνοχής. Η επόμενη διαφάνεια σας δείχνει ένα παράδειγμα. Πορτογαλία. Οι επιπτώσεις στο ΕΠ. Το βλέπετε στο πρώτο διάγραμμα. Και βλέπετε το επίπεδο όσον αφορά τις δαπάνες συνοχής 4% φτάνει το ΕΠ. Το 2007 και 2008. 4%. Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Τώρα η τεχνητή κατάσταση που πρέπει να απεικονίσουμε είναι με την υπόθεση ότι το 2009 σταματάει η συνοχή. Και το κάναμε λοιπόν με έναν τρόπο που δεν ήταν ο καλύτερος για μας, αλλά έπρεπε να το κάνουμε έτσι. Και θα έρθω μετά στο γιατί. Απασχόληση. Οι επιπτώσεις είναι μικρότερες από ό,τι στο ΕΠ. Γιατί η κύρια επίπτωση της συνοχής είναι παραγωγικότητα. Άρα έχετε λιγότερο κέρδος στην απασχόληση σε ποσοστά. Απορροφούνται λοιπόν τα κονδύλια. Το ισοζύγιο εμπορίου είναι αρνητικό όσον αφορά την παραγωγή αγαθών ε, κεφαλαίου, καταναλωτικά αγαθά. Και μετά την πάυση του προγράμματος, τότε έχουμε θετικές επιπτώσεις. Το επόμενο διάγραμμα δείχνει κάτι αντίστοιχο για την Πολωνία αυτή τη φορά. Εδώ η χρηματοδότηση ξεκινάει βέβαια το 2004 μετά την προσχώρηση της χώρας και αντίστοιχα βλέπετε τις επιπτώσεις στην, ε, στο ΕΠ, στην απασχόληση και στο εμπόριο. Εδώ βέβαια οι επιπτώσεις είναι μικρότερες γιατί είναι μικρότερο το διάστημα από ό,τι ήταν στην Πορτογαλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Εδώ λοιπόν βλέπετε το ΕΠΕ πρώτα απ' όλα, την απασχόληση όπως είπαμε και το ισοζύγιο εμπορίου. Μην πω σε λεπτομέρειες, πάντως αυτά σας δείχνουν πώ τα διαφορετικά ταμεία βελτιώνουν την απόδοση των δικαιούχων χωρών. Βέβαια, τα ποσά που παίρνουν οι χώρε είναι πολύ διαφορετικά. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε αυτέ τι επιπτώσει και να πούμε τα ιδιωτικά ταμεία είναι πιο αποτελεσματικά, για παράδειγμα, στην Πορτογαλία από ότι στην ε, Πολωνία. Η Πορτογαλία πήρε πολύ περισσότερα χρήματα κατά τη διάρκεια τη περίοδου από ότι η Πολωνία. Χρησιμοποιούμε γι' αυτό ένα μέτρο cumulative multiplier, έναν συσσωρευτικό πολλαπλασιαστή για να δούμε ποια είναι η απόδοση της επένδυσης. Άρα δεν εξαρτάται από την επένδυση ακριβώς που κάνατε, αλλά από την απόδοση αυτής της επένδυσης. Αν δείτε λοιπόν το επόμενο διάγραμμα θα δείτε πώς αυτός ο δείχτης ερμηνεύεται στην περίπτωση της Πολωνίας. Θα λέγαμε ότι ήταν είναι κινησιακού τύπου πολλαπλασιαστές αυτοί που χρησιμοποιούνται εδώ. Προχωρώντας τα χρόνια, τα κονδύλια τα οποία έρχονται στη χώρα αυξάνονται. Αυτός ο δείκτης αυξάνει, αυξάνει, αυξάνει και το 2020 βλέπετε ότι βρίσκεται στο 2,5. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ευρώ που παίρνετε έχετε 2,5 ευρώ επιστροφή σε όρους ΑΕΠ. Και στο επόμενο διάγραμμα βλέπετε το ίδιο αναχώρα. Οπότε βλέπετε πόσο αποδίδει η συνοχή στις διάφορες χώρες. Αριστερά έχετε την Ιρλανδία, καλύτερη απόδοση. Και μετά βέβαια υπάρχουν μικρές διαφορές. Εντάξει, η Λετωνία είναι δεξιά-δεξιά, αλλά δεν σημαίνει ότι η διαφορά είναι τόσο μεγάλη, απλώς είναι μικρότερη απόδοση. Γιατί είναι διαφορετική αυτή η απόδοση. Αυτό θα μας έβαζε βέβαια σε βαθιά νερά. Πρώτα απ' όλα έχει να κάνει με τη διάφρωση των οικονομιών των χωρών αυτών. Αν δείτε τις τρεις βαλτικές χώρες, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία, η Εστονία, Λιθουανία και Λετωνία με τη σειρά, σειρά μείωση. Ένας από τους λόγους είναι ότι η μεταποίηση στη Λετωνία είναι μικρότερη από τις στις τρεις βαλτικές χώρες. Αν λοιπόν ξεκινήσετε από το 2004 με τις τρεις αυτές οικονομίες των βαλτικών χωρών που κανονικά μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν όμως παρόλα αυτά διαφορές όσον αφορά στην ε, μεταποίηση. Θα περίμενε κανείς η οικονομία να ξεκινήσει με τις μικρότερες ε, επιπτώσεις. Και πράγματι αυτό βλέπουμε. Μπορούμε επίσης να συγκρίνουμε την Ιρλανδία με την Ελλάδα. Η διαφορά μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλη, αλλά και εδώ ισχύει το ότι ο μεταπηρικός τομέας ε, στην Ελλάδα είναι πολύ διαφορετικός ποιοτικά από ό,τι στην Ιρλανδία. Στην Ιρλανδία ο προσανατολισμός είναι περισσότερο εξαγωγές. Οπότε, τι περιμένετε να γίνει όταν σταματήσει η συνοχή, να πληγεί η Ιρλανδική οικονομία περισσότερο από ό,τι η ελληνική. Και όντως αυτό είναι και το συμπέρασμά μας. Εδώ βέβαια δεν πρόκειται για κανένα διαγωνισμό. Δεν θέλουμε να πούμε εδώ ότι αυτή η χώρα είναι καλή, η άλλη είναι κακή. Όσον αφορά το σχεδιασμό απορρόφησης των κονδυλίων, δεν είναι αυτό ο στόχος μας. Απλώ σα λέμε ποια είναι η κατάσταση όσο απορροφάνε κονδύλια συνοχή σε διάφορε χώρε. Προσπαθούμε τώρα να εκφράσουμε, είπαμε, ποσοτικά και τι επιπτώσει στι χώρε δωρητέ. Και εδώ πάλι χρησιμοποιούμε οικονομικά μοντέλα περιλαμβάνουμε και τις 27 χώρες, πλην 2, Βουλγαρία και Ρουμανία. Και εδώ κάνουμε προσωμείωση των επιπτώσεων ε, για την περίοδο 2000-2008. Κάνουμε επίσης προσημείωση όσον αφορά τα εμπορικά στοιχεία από τις χώρες δικαιούχους. Και συνδυάζουμε αυτές τις δύο προσωμιώσεις. Και έτσι βρίσκουμε το τελικό αποτέλεσμα, το καθαρό, αν είναι θετικό ή αρνητικό. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι ότι οι χώρες ε, δωρητές είναι πολύ βασικό κατά πόσο έχουν προσανατολισμό εξαγωγών ή όχι προς τις χώρες δικαιούχους. Η Γερμανία είναι εκείνη που έχει τον ε, πιο ψηλό τέτοιο προσανατολισμό προς τις χώρες δικαιούχους. Το 1 πέμπτο των εξαγωγών της Γερμανίας πάει προς τις χώρες δικαιούχους. Θα περίμενε κανείς η Γερμανία να υποφελείται πολύ. Λουξεμβούργο και κάτω χώρες έχουν χαμηλό τέτοιο προσανατολισμό εξαγωγών προς τις χώρες δικαιούχους. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά, ένα φίλτρο το οποίο θα επηρεάσει το αποτέλεσμα. Από την άλλη μεριά όμως οι χώρες δικαιούχοι εξάγουν επίση προς τις χώρες δωρητέ. Και εδώ Ισπανία και Πολωνία βλέπουμε ότι έχει τον πιο ψηλό προσανατολισμό εξαγωγών προς τις χώρες δωρητέ. 70% περίπου των εξαγωγών τους πάει προ τις χώρες αυτές. Στην περίπτωση της Ισπανία αυτό κυριαρχείται και στη Γαλλία πάει περισσότερε ε, εξαγωγέ. από την Πολωνία πάνε στη Γερμανία οι περισσότερες εξαγωγές τους και όσον αφορά τη Λετωνία και την Λιθουανία έχουν τον χαμηλότερο προσανατολισμό εξαγωγών προ τι χώρε δικαιούχου. Ίσως γιατί οι χώρε αυτέ, ε, όσον αφορά το εμπόριό του, εξαρτώνται ακόμα σε ένα μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία. Μειώνεται η σχέση αυτή, αλλά όσον αν εξακολουθεί να υπάρχει. Εξάγω στη Ρωσία, όχι στις χώρε δικαιούχου τόσο. Βλέπουμε εδώ πέρα το αποτέλεσμα. Γαλλία, παράδειγμα τη Γαλλία. Η Γαλλία έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα, εμπορικά πλεονεκτήματα που φαίνονται εδώ. Και φαίνονται πολύ ωραία και θετικά και τα λοιπά. Τελικά όμως δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Απ' την άλλη μεριά όμως, στη Γερμανία βλέπουμε στην αρχή αρνητικές επιπτώσεις επειδή ακριβώς συνεισφέρει λοιπά. Όταν το 2008 σταματάει η συνοχή, τότε ξεκινάει το θετικό αποτέλεσμα, το θετικό ισοζύγιο. Μεγάλη διαφορά λοιπόν ανάμεσα σε δύο χώρες καθαρούς δωρετές. Μετά έχουμε τις κάτω χώρες. Είδαμε ότι είναι χώρα η οποία είχε πολύ χαμηλό προσανατολισμό εξαγωγών προς τις δικαιούχους χώρες. Εδώ βλέπετε ότι οι επιπτώσεις ε, στο ΕΠΟ είναι μεγάλες, αρνητικές, 1% φτάνουν και ο λόγος είναι ότι οι κάτω χώρες παίρνει όλο αυτό το βάρος της εισφοράς της χωρίς εμπορικά να υποφελείται τόσο. Μετά όμως αλλάζει η κατάσταση μετά το 2009-2010 και υποφελείται από τις εμπορικές συναλλαγές και η Ολλανδία. Υπάρχει μεγάλη διαφορά λοιπόν ανάμεσα στις χώρες. Τι συμπέρασμα μπορεί να βγάλει κανείς όσον αφορά τις επιπτώσεις στις χώρες δικαιούχους. Οτιδήποτε σταματάει 31 Δεκεμβρίου 2008 το ρολόι του υπολογισμού σφάλει. Γιατί βλέπετε κι εσείς ότι οι επιπτώσεις προχωράνε. Πρέπει να συνεχίσει κανείς την ανάλυση και μετά την προγραμματική περίοδο για να καταλάβει τις πραγματικές επιπτώσεις. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς. Οι επιστροφές, η απόδοση των ε, δαπανών συνοχής διαφέρουν από χώρα σε χώρα εξαιτία διαρθρωτικών διαφορών στις οικονομίες. Όμως μπορεί αυτό να οφείλεται και στην αποτελεσματικότητα και την απόδοση της ίδιας της πολιτικής ε, συνοχής βάσει του εθνικού σχεδιασμού και της εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν ποιοτικέ διαφορές. Εμείς εκφράσαμε ποσοτικά την κατάσταση, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να δούμε ποιος τελικά σχεδιάζει την ε, συνοχή και πώς την εφαρμόζει. Ποιος το, κάνει το σχεδιασμό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ποιος με λιγότερο καλό τρόπο. Ποιος ε, εφαρμόζει στην πράξη τη συνοχή καλύτερα και ποιος λιγότερο καλά. Έτσι κι αλλιώς οι διαδικασίες είναι περίπλοκες όπως ξέρουμε. Τώρα οι δαπάνες συνοχής Ε, αυξάνει και τη ζήτηση για εισαγωγές από τις δικαιούχους χώρες. Η ζήτηση για εισαγωγέ παραμένει υψηλή και μετά την περίοδο εφαρμογή τη συνοχή. Το εμπορικό ισοζύγιο γίνεται θετικό. Δηλαδή, μία από τις επιπτώσεις απορρόφησης κονδυλίων συνοχής και καλής τους χρησιμοποίησης είναι ότι ο προσανατολισμός για εξαγωγές αυξάνει και γίνεται πιο ανταγωνιστικό σε διεθνές επίπεδο. Ο προσανατολισμός τώρα των χωρών που συνεισφέρουν περισσότερο στο εμπόριο με τις χώρες δικαιούχους επηρεάζει και την μεταφορά του ισοζυγίου στο εμπόριο. Μπορεί βέβαια να υπάρχουν και ιστορικοί λόγοι. Οι επιπτώσεις τώρα στο ΕΠ για τη χρηματοδότηση είναι κατερνητικό σε όλες τις περιπτώσεις. Στη Γερμανία μερικές φορές υπάρχει διαφοροποίηση στα κρατήδια της Τέσσερα Ανατολικής Γερμανίας. Οι επιπτώσεις τώρα στους ε, δωρητές, το ΕΠ των δωρητών από τους δικαιούχους. Είναι θετικό για το ισοζύγιο το εμπορικό. Επηρεάζεται βέβαια από τον εμπορικό προσανατολισμό. Με εξαίρεση είπαμε τις βαλτικές χώρες επειδή έχουν τις συναλλαγές ακόμα με τη Ρωσία. Εξαρτάται από τις εμπορικές συναλλαγές που έχουν οι χώρες φορής με τις δικαιούχους χώρες. Για την απασχόληση στις χώρες δωρητές, οι επιπτώσεις είναι όπως και για το ΕΠ, αλλά κάπως μικρότερες σε κλίμακα. Το μέγεθος των επιπτώσεων πάντως είναι σχετικά περιορισμένο αν δούμε τη συνεισφορά στο προπολογισμό. Η Γερμανία συνεισφέρει μισό της εκατό χαμηλότερα στο ΕΠ. όσο για τις δαπάνες μπορεί να είναι στο 40% του ΕΠ. Η συνεισφορά τώρα στον προπολογισμό για τη συνοχή εννοείται ότι ευνοεί το ισοζύγιο. Οι επιπτώσεις τώρα στο δημόσιο τομέα. Είναι αρνητικό κατά την περίοδο εφαρμογής, αλλά θετικό μετά την εφαρμογή της συνοχής. Και αυτό έχει να κάνει με το ότι είσαστε καθαρό εισφορέα. Οι επιπτώσεις τώρα στην αποδοτικότητα και στο cash flow των καθαρών δωρητών επίσης είναι αρνητικό κατά τη διάρκεια τη συνοχή και θετικό μετά. Πάλι γιατί πρόκειται για καθαρό εισφορέα που πλήττεται. Τι γίνεται τώρα με τις ε, μικροεπιπτώσεις με συμβάσεις από τις χώρες δωρητές. Όταν εξετάζουμε αυτό το θέμα, διαπιστώνουμε ότι από τις χώρες δωρητές έχουν ε, πολλές φορές υποσυμβάσεις, εργολαβίες δηλαδή, με χώρες δικαιούχους. Κάτι που είναι αρκετά περίπλοκο και όχι πάντα πολύ καθαρό. Οι έρευνες σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που κάναμε έδειξαν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν έχουν συλλεχθεί στοιχεία καθόλου για την ε, δημοσιονομική περίοδο 2000-2006. Κάτι το οποίο μας εξέπληξε. Οπότε δεν μπορούμε εδώ να δώσουμε καμία αξιόπιστη απάντηση σε αυτό το ζήτημα. Για δύο λόγους. Ένα είναι ότι είναι έτσι κι αλλιώς περίπλοκο ζήτημα. Δεν είναι καθόλου απλό. Και δεύτερον, γιατί κανείς δεν ασχολήθηκε να συλλέξει δεδομένα γι' αυτό. Μπορεί να υπάρχουν πολύ καλοί λόγοι. Είναι θέμα απορρίτου εμπορικού ίσως. Είναι θέμα έλλειψης επιθυμίας της Κομισιόν να αναμειχθεί σε αυτό το επίπεδο. Το αποτέλεσμα πάντως είναι ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε σε μικρό επίπεδο τι έγινε. Για να ολοκληρώσω κάποιες συστάσεις. Η ανάλυση μας βασίζεται σε στοιχεία της ανάλυσης κόστος-κέρδος. Διαπιστώσαμε ότι ελάχιστα από αυτά έγιναν γνωστά. Και οι τρεις έχουμε δουλέψει πολύ σε αυτό το τομέα για πολλά χρόνια και όμως ποτέ, μα ποτέ δεν είδαμε δημοσίευση μια τέτοιας ανάλυσης κόστους κόστους-οφέλους. Ε, και είναι κρίμα. Συνεχίζεται αυτή η κατάσταση τι να κάνουμε, είναι παρενέργεια ας πούμε. Τη αποσύρει λοιπόν τέτοιων μελετών είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε επιχειρήματα που χρειάζονται για να αξιολογήσουμε το κατά πόσο οι χώρες σχεδιάζουν και εφαρμόζουν καλά την πολιτική συνοχής. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι επειδή εμεί περιοριστήκαμε μόνο στη συνοχή, ήταν όντω αυτό κάτι που μας περιόρισε. Γιατί θέλαμε περισσότερο να το στιάσουμε με την εσωτερική αγορά, με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, ευρώ. Όμως αυτοί οι παράμετροι αλλάζουν το κλίμα μέσα στο οποίο οι χώρες λειτουργούν. Και πολλές φορές ευνούν τα κέρδη κάποιων χωρών που καταφέρουν καλύτερα να τα βγάλουν πέρα μέσα στην ευρωπαϊκή αγορά. Τέλος, μας ζητήθηκε να κοιτάξουμε την περίοδο 2000-2006. Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιρλανδία εποφελήθηκαν από την πολιτική συνοχής από το 1989. Μα ζητήθηκε λοιπόν τεχνητά κάπως να το δούμε και αυτό. Παρόλο που η δουλειά στις χώρες αυτές συνεχίζεται με κάποιες μικρές αλλαγές στα προηγούμενα προγράμματα. Για την περίοδο 2007-2013 θα δούμε τι έχει γίνει στις νέες χώρες, μια που περνάνε από την πρώτη τους ε, περίοδο 2006, με 2006, στη δεύτερη 2007 με 2013. Τα προγράμματα τους αυτά θα πρέπει συσσωρευτικά να αναλυθούν και όχι να τα χωρίσουμε διοικητικά γιατί αυτό είναι ένας πολύ τεχνητός τρόπος. Ελπίζουμε ότι θα έχετε την ευκαιρία να κοιτάξετε τη δουλειά μας λεπτομερέστερα, αλλά συνοπτικά κάπως αυτό είναι που κάναμε. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να συζητήσουμε τώρα τα της παρουσιάσεως. Yes, Ένα ερώτημα. Ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσίασή σας. Άκρως ενδιαφέρουσα. Γνωρίζετε ότι η πολιτική συνοχής επί του παρόντος ε, δεν ε, πάει τόσο καλά δεν προωθείται σωστά εντός, των, εντός του θεσμικού μας οργάνου και θέλουμε να έχουμε τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες. Θέλουμε να ξέρουμε τη σχέση κόστους-οφέλους της πολιτικής αυτής. Μας λέτε ότι δεν έχετε αριθμητικά στοιχεία που μας επιτρέπουν μία ανάλυση τέτοια κόστους-οφέλους. Ποιος έχει τις πληροφορίες και πώς κατά την άποψή σας μπορούμε να αποκτήσουμε τις εν λόγω πληροφορίες Ποιος είναι ο που διαθέτει αυτές τις πληροφορίες και που θα μπορούσε να μας βοηθήσει. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό σήμερα να πετύχουμε διαφάνεια όσον αφορά αυτά τα στοιχεία. Τα αναλυτικά στοιχεία που είναι πολύ ουσιαστικά. Πέρα από την άμεση παρέμβαση των ευρωπαϊκών πόρων στην επικράτειά μας, η έμεση ε, συνέπεια, ο έμεσος αντίκτυπος έχει σημασία επίσης περνάμε κρίση, όλα τα στοιχεία είναι σημαντικά. Πώς μπορούμε λοιπόν να σας βοηθήσουμε για να αποκτήσετε από κάποια από τα θεσμικά μας όργανα αυτά τα στοιχεία. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ε, Ποιος θα δώσει απάντηση. Έχει το λόγο καθηγητά. Φίξατε δύο σημαντικά θέματα. Αφενός τον τρόπο που γίνεται η ανάλυση κόστους-οφέλους και το άλλο, πώς μπορεί να πει κανείς ήδη από τώρα, από σήμερα κάτι σχετικά με τη συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων μέσα στην κρίση και ποια θα είναι η επίδραση αυτής της ε, συμβολής. Για το δεύτερο θα πει ο συναδελφός μου κάτι για τις αναλύσεις κόστους-οφέλους προκαταρκτικά, δηλαδή πριν από την εφαρμογή μεγάλων έργων, αυτές είναι υποχρεωτικές για έργα που είναι παραπάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές γίνονται αυτομάτως τότε. Η αξιολόγηση γίνεται μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενδεχομένως με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την αξιολόγηση και στη βάση αυτής της ανάλυσης κόστους κόστος-οφέλους λαμβάνει τη τελική απόφαση για το έργο. Πρόσβαση σε αυτές τις αναλύσεις κόστος οφέλου στην πραγματικότητα δεν έχουμε. Δεν είναι δηλαδή ε, δεν δημοσιοποιούνται δηλαδή. Μόνον εφόσον δημοσιευτούν μπορεί κανείς να κρίνει ποιες είναι οι επιπτώσεις της ανάλυση κόστου ωφέλους για την έγκριση του έργου ή, εν πάση περιπτώσει, ποια, ποιο κόστος και ποια ωφέλη θα προέκυπταν από την υλοποίηση ή μη του έργου. Όσο δεν έχει δημοσιευτεί αυτή η ανάλυση κόστου ωφέλους, δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά τα πράγματα. Ωστόσο υπάρχουν οι αναλύσεις αυτές για τα μεγάλα έργα. Τώρα, ποιε διαδικασίες πρέπει να τηρούνται, δεν μπορώ να σας το πω. Αυτά είναι οργανωτικά διαδικαστικά τεχνικά θέματα τα οποία θα πρέπει να διασαφίζει το Κοινοβούλιο σε συνεργασία με τις διοικητικές αρχές. Όμως, επαναλαμβάνω, υπάρχουν οι αναλύσεις κόστους ωφέλους για τα μεγάλα έργα. Από την άλλη μεριά, είναι ενδιαφέρον να δει κανείς ότι μέτρα τα οποία σχεδιάζονται για να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις κοινωνικές και στην απασχόληση για παράδειγμα στην ε, Ιρλανδία έγινε μέσα στα πλαίσια μιας midterm review, μιας ενδιάμεσης επανεξέτασης και στη Γερμανία επίσης έγιναν κάποιες αξιολογήσεις για την ανάπτυξη. Πάλι αυτά όμως δεν είναι στάνταρτ, αυτά χρησιμοποιούνται κάπου κάπου γίνονται εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να έχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τις επιπτώσεις και κοινωνικές αλλά και στην απασχόληση. Αυτά για ε, την ανάλυση, τις αναλύσεις μάλλον κόστους ωφέλους και ίσως ο Τζον μπορεί να πει λίγα πράγματα για τις επιπτώσεις της κρίσης. Άνθρωποι όπως εσείς οι βουλευτές όταν εξετάζουν την πολιτική συνοχής προσπαθούν να σταθμίσουν διοικητική, επιπλοκή και περιπλοκή και οικονομικά, οικονομικές πτυχές. Ποιο είναι το πρόβλημα. Όπως προαναφέρθηκε, κάποιοι από τους κανόνες που διέπουν τα διοικητικά των διεθνωτικών ταμείων έχουν περιπλακεί τόσο που οι εθνικές κυβερνήσεις και οι περιφέρειες κινούνται προς προγράμματα που είναι εύκολο να περάσουν το σύστημα περισσότερο παρά προς τα προγράμματα εκείνα που είναι πιο επωφελή οικονομικά. Από την άλλη πλευρά εμείς οι οικονομολόγοι τα βλέπουμε διαφορετικά. Και τι είναι ενδιαφέρον ότι δύο σημαντικές υποθέσεις όπου η γέννη και προσπάθεια για να είμαστε ομά ειλικρινείς όσον αφορά ενδιάμεση αναθεώρηση για να δούμε πού η διοικητική μέρη ήταν αποτελεσματική και πού να σταματήσουν τα προγράμματα. Ήταν η Ιρλανδία και η Γερμανία. Εκεί υπήρξε συνεργασία. Και μια κυβέρνηση κατάλαβε ότι έπρεπε να γίνει ιδέουσα προσπάθεια. Αν θεσπίσει νόμους η Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες αυτή δεν θα είναι τόσο ανοιχτή. Διότι μια χώρα έκανε ένα είδος αυτοανάλυσης. Σε διεθνή βήματα παρισφρίουν άλλοι παράγοντες. Αν εγώ είμαι ομά ειλικρινής για τα που σπαταλήθηκαν χρήματα στην Ιρλανδία, μπορεί να τα πάρουν από μένα και να τα δώσουν σε μια άλλη χώρα η οποία δεν είχε την ίδια ειλικρίνεια με την Ιρλανδία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτά παίζουν ρόλο. Μπορεί να το επιβιώσει και ο καθηγητής Ζαλέσκης ο την Πολωνία. Ε, είναι πάρα πολύ περίπλοκα τα πράγματα και έτσι δεν τίθεται τα σωστά ερωτήματα. Δηλαδή ο Ευρωπαίος φορολογούμενος στις ε, ε, χώρες παίρνει πίσω τα λεφτά του, πετυχαίνει τα αποτελέσματα τα ευκταία. Δεν ξέρω, ίσως ο καθηγητής Ζαλέσκη θέλει να πει κάτι πάνω σε αυτό. Ευχαριστώ. Αν επιτρέπετε θα ήθελα να επιβεβαιώσω πράγματι ότι οι διοικητικοί κανόνες είναι περιπλοκότατοι όσον αφορά την πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους σε χώρες κυρίως όπως είναι η Πολωνία που η Πολωνία εδώ και μερικά χρόνια μπορεί να ωφελείται από τους ευρωπαϊκούς πόρους. Το πιο σημαντικό τώρα είναι η απορρόφηση των πόρων. Η αποτελεσματικότητα δεν είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Γιατί, πώς δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση. Η πρόσβαση στα ταμεία, στους πόρους, ε, περιορίζεται από πληθώρα συνθήκων και όρων. Και έχει γίνει κατάσταση τόσο περίπλοκη που ακόμα και οι κρατικοί φορείς δεν γνωρίζουν όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται. Άρα ε, προωθούμε προγράμματα που θεωρούμε ότι σίγουρα θα ωφεληθούν από τους αναγκαίους πόρους. Δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε κάτι που θεωρούμε ότι είναι αρκετά παρακινδυνευμένο λόγω της μεγάλης περιπλοκότητας των κανόνων που επιβάλλονται. Αυτά συνεπάγονται μεγάλα ποσά που δίδονται, αλλά υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβαση ποσούς. Στα ποσά, συγγνώμη. Προσπαθήσαμε να αναλύσουμε την κατάσταση όσον αφορά τις συμβάσεις που συνάπτουν οι ξένες εταιρείες. Απλώς για στατιστικούς σκοπούς κάνουμε την όλη προσπάθεια. 14% των συμβάσεων, 14% κατά την περίοδο προγραμματισμού που συζητούμε, το 14% λοιπόν των προγραμμάτων αφορούσε συμβάσεις από τις οποίες ωφελήθηκαν οι εταιρείε των χωρών δωρητών. Όσον αφορά την ερμηνεία, όπως είπε ο Τζον, είδαμε όπου σε πολλές συμβάσεις την υπεργολαβία ανέλαμβαναν ε, πολωνικές ε, εταιρείες. Μπορεί να μηνεθούν ποικίλω αυτά τα στοιχεία. Υπάρχουν όμιλοι επιχειρήσεων όπου το πολωνικό κεφάλαιο είναι παρόν. Άρα είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει κανείς αν πρόκειται για σύμβαση που αφορά αποκλειστικά μια ξένη εταιρεία ή ε, ένα κράμα εταιρεών. Αυτό το 14% είναι ένας δείκτης, αλλά είναι αβέβαιος δείκτης, δεν είναι απόλυτος δείκτης, ίσως. Ε, υπάρχει και άλλο ένα στοιχείο που αφορά την ε, ανάλυση κόστους-οφέλους. Στην περίπτωση μεγάλων προγραμμάτων όπου το συνολικό ποσό ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ μπορεί κανείς να έχει μία πρόσβαση σε τέτοια ανάλυση κόστους ωφέλους. Αλλά υπάρχουν πολλά προγράμματα που ξεπερνούν ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυτό το ποσό. Άρα θα έπρεπε να γίνεται αναλυτική μελέτη σε επίπεδο μακροοικονομικό και μικροοικονομικό για να ληφθούν υπόψη αυτά τα στοιχεία. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, να μαζέψουμε τέτοια στοιχεία. Η συλλογή στοιχείων ανάμεσα στο μακρο και μικροοικονομικό επίπεδο θα ήταν κρίσιμη σημασία. Ο Τζον και ο Γκεράρ το έκαναν αυτό εν μέρη κατά το παρελθόν και δυστυχώς τέτοιες μελέτες δεν υλοποιήθηκαν πραγματοποιηθήκαν σε όλες τις μελέτες. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Ε, καταρχήν ήθελα να κάνω μια πρόταση. Δεν ξέρω πόσο αυτό αφορά και τους υπόλοιπους συναδέλφους, αλλά εμένα με αφορά. Ε, νομίζω ότι η μελέτη ήταν πολύ σημαντική. Ε, χρειάζεται να μελετήσουμε λίγο παραπάνω, να δούμε και διάφορες πλευρές που αυτή τη στιγμή όταν πρωτοβλέψαν τόσο σημαντικό πράγμα ε, δεν έχει το καιρό να τα αφομοιώσει και ενδεχομένω ε, να επανέλθουμε, Είμαι σίγουρο ότι θα έχουμε όλοι και περισσότερε ερωτήσει ώστε να ε, είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει με τα σημερινά, καταρχήν. Ε, νομίζω ότι θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε τους ε, μελετητές μας να ερευνήσουν λίγο περισσότερο αυτό το ζήτημα με τι συμβάσει, το οποίο έγινε λόγος και εισηγητικά αλλά και τώρα ακούστηκε μια άποψη. Γιατί βεβαίως το 14% μπορεί να είναι μικρό, μεγάλο ε, σαν αριθμό, αλλά έχει μια σημασία να δει κανεί και λέω για το 14% που τουλάχιστον αυτό είναι κάπως συγκεκριμένο, ε, έχει μια σημασία και το τι οικονομικό μέγεθος είναι το 14%. Γιατί μπορεί να είναι ο αριθμός των συμβάσεων σχετικά μικρός, αλλά είναι, αν είναι όμως το μεγάλο μέρος των ποσών, αλλάζουν τα πράγματα. Ένα δεύτερο ζήτημα ε, σημαντικό νομίζω και από άποψη πολιτικής είναι τελικά και ξέρετε ε, θέλω να εκφράσω έτσι λίγο μια άποψη από μια χώρα όπως η Ελλάδα που είχε ε, τα αποτελέσματα που είχε που δείχνει η μελέτη τελικά φαίνεται ότι και οι δωρητές χώρες έχουν όφελος από τα ταμεία συνοχής και όχι μόνο οι χώρες που δέχονται. Γιατί η επικρατούσα άποψη είναι ότι τελικά οι δωρητές χώρες χάνουν και οι χώρες που δέχονται κερδίζουν. Από τη μελέτη και αν είναι σωστά νομίζω ότι τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. Και αυτό είναι σημαντικό ε, για να είναι γνωστό στους ε, ε, λαούς της Ευρώπης. Τρίτο ζήτημα. Μιλάμε για συνοχή. Ποιο είναι το κριτήριο. Πότε μπορεί να πει κανείς ότι μια πολιτική συνοχή είναι καλή ή δεν είναι καλή. Μας είπαν εδώ ε, οι κύριοι και σωστά ε, στοιχεία με ΑΕΠ, με απασχόληση κτλ. Μήπως πρέπει να βρεθεί ένα άλλο κριτήριο. Παραδείγματο χάρη, τη συνοχή γιατί τη θέλουμε, τη θέλουμε ώστε το επίπεδο ανάπτυξη να είναι περίπου το ίδιο, φαντάζομαι. Έτσι. Ε, Μήπω θα έπρεπε να δούμε το στοιχείο τη παραγωγικότητα τη εργασία, πόσο αυτό ανεβαίνει, πόσο τα μία συνοχή συμβάλλουν σε αυτό, ώστε πράγματι να έχει μια συνοχή. Και τελευταίο, θα ήθελα να κάνω την εξή ερώτηση. Μα είπε η μελέτη, μα είπαν ε, οι κύριοι που παρουσιάσαμε, ότι περίπου 50% των προγραμμάτων πήγαν στις υποδομές, 36% στους ανθρώπινους πόρους και 16% μόνον στον παραγωγικό τομέα. Έχουν τη γνώμη ότι αυτές είναι οι καλές αναλογίες για τις χώρες της συνοχής. Ε, μήπως πρέπει εκεί, δεν λέω τώρα, το δούμε, το μελετήσουμε μελλοντικά, να υπέλθουν κάποιες αλλαγές ώστε τα αποτελέσματα να είναι πιο αποτελεσματικά, ώστε να γίνει πιο γρήγορα η συνοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Professor Lundit, would you reply to these questions, please? Μπορείτε να απαντήσετε, αν θέλει κάποιος, εσείς. παρουσιάσαμε τα αποτελέσματά μας αναχώρα και δείχνουμε ότι σε μια χώρα όπως η Ελλάδα η συνοχή έχει καλύτερο αποτέλεσμα στους μακροοικονομικούς δείκτες. Εμείς το ερμηνεύουμε αυτό λέγοντας ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα συγκεκριμένα, η συνοχή αποδίδει. Αυτό όμως είναι μερική μέτρηση της συνοχής, όπως είπατε και εσείς. Η συνοχή είναι μια έννοια η οποία καλύπτει όλες τις χώρες μέλη της Ένωσης και έχει το νόημα να αποφευθεί μια δημιουργία μιας Ευρώπης με χαμένους και κερδισμένους. Έχει μια διάσταση η οποία ξεπερνά ε, απλώς την οικονομική αποδοτικότητα. Δηλαδή ακόμα και αν δείχνουμε ότι το κόστος για τις καθαρές συνεισφέρουσες χώρες δεν εξισορροπεί ακριβώς την ωφέλεια για τις απολύπτριες χώρες. Δηλαδή δεν υπάρχει εν τέλει καθαρό κέρδος για την Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά η πολιτική συνοχή μπορεί να θεωρηθεί κάτι τίτο θετικό γιατί έχει και μια ευρύτερη διάσταση της συνοχής για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Αυτό είναι σημαντικό, πρέπει να τονιστεί. Αν βγούμε λιγάκι τώρα έξω από τα στενά όρια του μας. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η πολιτική συνοχή από τότε που διευρύνθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 80 έχει την τάση να ενισχύσει περισσότερο την εθνική συνοχή αλλά την περιφερειακή διαφοροποίηση. Αυτό φαίνεται και από την εθνική βιβλιογραφία. Υπάρχει το ελαφρώς παράδοξο παίρνοντας για παράδειγμα την Πολωνία. Στο σύνολό της η Πολωνία προχωρεί με αρκετά καλή ταχύτητα προς κάποιο επίπεδο κατά να ΕΠ κοντά στο μέσο όρο της, ε, της Ένωσης, αλλά οι περιφέρειες, οι πολωνικές περιφέρειες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλες ακολουθούν στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό βέβαια θέτει ένα ευρύτατο θέμα για το πώς αντιμετωπίζοντας μια τέτοια εξέλιξη θα πρέπει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για πρόβλημα που νομίζω μάλλον πρέπει να συζητηθεί στο Κοινοβούλιο και λιγότερο μεταξύ των οικονομολόγων. Κατά μία έννοια, αν και ορισμένες περιφέρειες μέσα σε μια χώρα εποφελούνται περισσότερο από άλλες περιφέρειες μέσα στην ίδια χώρα, αυτές που αναπτύσσονται αργότερα, παρόλα αυτά εποφελούνται αφού άλλωστε ενισχύεται κάποια μεταναστευτική ροή από τις περιφέρειες αυτές προς άλλες περιφέρειες. Καθαρό παράδειγμα η Ιρλανδία με μετακίνηση πληθυσμών από το φτωχότερο νότο και δύση προς το κέντρο και την ανατολικό μέρος της χώρας που είναι το πλουσιότερο. Σε ό,τι αφορά την κατανομή των πόρων μεταξύ υποδομής, ανθρώπινου δυναμικού κλπ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα τα τελευταία 20 χρόνια στην Ευρώπη. Εγώ ήμουν από την αρχή του σχεδιασμού των διαρθωτικών ταμείων για την Ιρλανδία, το 1993 ήδη, όταν η Ιρλανδική κυβέρνηση ζητούσε 45% συνολικά των χρημάτων να δοθεί στο ανθρώπινο δυναμικό. Και ανέκραξε με τρόμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτά πράγματα δεν γίνονται. Νομίζω τελικά καταλήξαμε να δαπανίσουμε 35% για το ανθρώπινο δυναμικό. Ταυτόχρονα η Πορτογαλία για ανθρώπινο δυναμικό έδωσε ένα ελάχιστο ποσοστό και τα περισσότερα αρχικά κεφάλαια τα διέθεσε στην ε, δημιουργία υποδομή. Και είδα εγώ τα ωφέλη που είχαν από αυτά με του καταπληκτικού αυτοκινητοδρόμου. Αυτά είναι επιλογέ αναχώρα. Δεν ε, γίνονται πάντοτε με τον πιο λογικό τρόπο. Καμιά φορά απηχεί κάποιες προτεραιότητες οι οποίες ξεπερνούν και τα καθαρά οικονομικά δεδομένα. Δεν υπάρχουν και μαγικές λύσεις άλλωστε. Μερικές χώρες με την υποδομή συνδέουν τι αγορέ τους με τις κεντρικές ευρωπαϊκές αγορές και αυτό είναι σημαντικό. Για τι νέες χώρες μέλη είναι σαφές ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, το κεντρικό στατιστικό μα γραφείο έκανε μια μελέτη τελευταία για ε, τα μεταναστευτικά ρεύματα που έρχονται στην Ιρλανδία από Λιθουανία και Πολωνία και ο μέσος όρος της εκπαίδευσης των μεταναστών ήταν πολύ ψηλότερο από το μέσον όρο των Ιρλανδών εργατών. Άρα, σε αυτές τις ανατολικές χώρες και άλλες, το ανθρώπινο δυναμικό είναι υψηλό ε, δυναμικά κεφάλαιο. Από την άλλη μεριά έχουν όμως ε, καταραίουσα υποδομή από την παλαιά ε, κληρονομιά τους. Έχετε δίκιο λοιπόν σε αυτά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ποστινάρου. Ε, ε, Πρόεδρε, η μελέτη που μας παρουσιάστηκε είναι ευπρόσδεκτη. Είναι πολύ σχετική με το θέμα μας. Και είναι πολύ προχωρημένη σε κάποια σημεία. Εγώ σαν μη οικονομολόγος πρέπει να πω ότι μόνο οικονομική διάσταση και η παρουσίαση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη σχέση που υπάρχει μεταξύ χωρών δωρητριών και χωρών δικαιούχων μόνο αυτή η προσέγγιση είναι ατελής και μπορεί κάπου να δημιουργεί αντιφάσεις. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε μια πραγματικότητα που λησμονούν καμιά φορά οικονομολόγοι. Δεν είμαι οικονομολόγος εγώ. Αλλά τώρα καθυστερημένα διαβάζω ε, βιβλία για οικονομία. Είναι πολύ πιο περίπλοκη η σχέση μεταξύ χωρών δωρητριών και δικαιωχών χωρών. Δείχνουν κάποιε μελέτε ότι οι πολιτικέ συνοχή μπορεί να έχουν πάντα θετική συνέπεια και αποτέλεσμα win-win από ό,τι δείχνουν οι μελέτε αυτέ. Και είναι θέση οικονομολόγων αυτή, που είπαν ότι η πρώτη πραγματική οικονομική κρίση στις αρχές της δεκαετίας του 90 στις χώρες Δυτικής Ευρώπης θα μπορούσε να έχει αποφευθεί ακριβώς διότι η Ευρώπη επεκτάθηκε προς τα 10 νέα κράτη-μέλη και μετά στα 12 νέα κράτη-μέλη. Έτσι, οι ευρωπαϊκές οικονομίες της Δύσης μπόρεσαν να ωφεληθούν από αγορέ καινούριε. Και αυτός ήταν ένα παράγοντα ανάπτυξης. Αυτό δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε. Υπάρχουν ωφέλη και από τις δύο πλευρές. Ένα δεύτερο στοιχείο που θέλω να αναφέρω. Οι βασικοί οικονομικοί φορείς στις χώρες που δέχονται χρηματοδότηση από την πολιτική συνοχής, επαναλαμβάνω, αυτή η οικονομικοί φορείς, οι βασικοί οικονομικοί φορείς, ξεκινώντας από τις τράπεζες, επενδυτικά ταμεία κλπ, είναι φορείς όλοι αυτοί οι οποίοι είναι εταιρείε που έχουν κεφάλαιο και το κεφάλαιο αυτό προέρχεται από τις δωρήτριες χώρες ή θυγατρικές των εταιριών που βρίσκονται στις ε, χώρες δωρήτριες. Λοιπόν, αυτή είναι η συνέπεια win-win, όπου όλοι κερδίζουν. Τρίτο στοιχείο. Αν κοιτάξετε και δείτε ποια συστήματα ισχύουν όσον αφορά τις συμβάσεις. Οι βασικές συμβάσεις που συνάπτονται στις δικαιούχες χώρες συνάπτονται κυρίως όταν πρόκειται για μεγάλα έργα, μεγάλα ποσά και πολύ συχνά σε αυτές τις συμβάσεις αναμειγνύονται επιχειρήσεις ή θηγατρικές επιχειρήσεις κάποιων επιχειρήσεων που εν γέννη ε, προέρχονται από τις δωρήτριες χώρες. Οπότε ξανά έχουμε ένα αποτέλεσμα που όλοι κερδίζουν. Win-win. Δεν ισχύει πάντα αυτό, αλλά μερικέ φορέ ισχύει. Άλλο στοιχείο. Το τραπεζικό σύστημα δεν λαμβάνει υπόψη την πολιτική συνοχής βεβαίω, αλλά όλε οι δικαιούχε χώρε έχουν τραπεζικό σύστημα που ελέγχεται ή επηρεάζεται από τραπεζικά συστήματα που υπάρχουν στις ε, δωρήτρες χώρες. Σε, μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα στη στιγμή κρίσης αυτό, αλλά και αρνητικές συνέπειες, παραδείγματο χάρη κερδοσκοπία επί του εθνικού νομίσματος σε Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία. Από που συνδέονται με τις δωρήτριες χώρες. Όλα αυτά παίζουν ρόλο στην, ε, στην υπόθεση αυτή τη θεωρητική του win-win όπου όλοι κερδίζουν. Και τέλος, η διαδικασία μετεγκατάστασης κάποιων εταιριών που πάνε από τις δωρήτριες χώρες προς τις δικαιούχες χώρες και το κάνω αυτό γιατί την πιο χαμηλή μισθή μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις να κρατήσουν έτσι την ανταγωνιστικότητά τους και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και ε, στο τοπικό επίπεδο. Volkswagen και Skoda και Dacia και Renault. Η Renault χάρη στην Dacia της Ρουμανίας γνώρισε θεματική ανάπτυξη. Ακριβώς διότι μετεγκατάστηκε η Renault και πήγε στη Ρουμανία. Οπότε είχαμε διάφορα αποτελέσματα. Έλαβαν υπόψη χαμηλότερους μισθούς, χαμηλότερη φορολογία κλπ. Αυτές οι πτυχές δεν μπορούμε να τις λησμονούμε. Οπότε, η ανάπτυξη μέσω πολιτικής συνοχής, η μείωση της διαφοράς ανάπτυξης μεταξύ δωρητριών χωρών και δικαιούχων χωρών και ε, αποτελούν προϋποθέσεις για την επιβίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας όλες αυτές οι συνιστώσεις. Είναι η μόνη δυνατότητα να αποφύγουμε διαφορές, αποκλίσεις που εντός μιας κρίσεως θα μπορούσαν να συμβούν. Το υποστηρίζουν αυτό και τα στατιστικά στοιχεία και νομίζω τα δικά στατιστικά στοιχεία, η μελέτη σας, είναι μια πρόσκληση για να συνεχιστεί αυτή η πολιτική της συνοχής και δεν θα πρέπει να κάνουμε αλλαγές που θα μας οδηγήσει μόνο προς ανταγωνιστικότητα, προς συναγωνισμό που ε, μπορεί να αυξήσουν ε, τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών πιστεύω. Ευχαριστώ την προσοχή σας. Uh, Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έμαθα ότι οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί, οι Αυστριακοί καλά θα ήταν να διπλασιάσουν ή να τριπλασιάσουν τις εισφορές τους στη συνοχή και τότε τα πράγματα θα πάνε τρεις φορές καλύτερα για τους ίδιους. Αυτά είπατε με, λίγο, με λίγα λόγια. Τώρα, για τις μετακινήσεις Έχετε δίκιο, αλλά οι βιομηχανίε οι ε, οποίε πάνε έτσι κι αλλιώ στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στην Τσεχία, πάνε για λόγου δικού του οικονομικού. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να τους δίνονται από πάνω και ευρωπαϊκά κονδύλια. Για τι ε, μετακινήσεις εδρών επιχειρήσεων και εμείς αλλά και οι Γάλλοι είμαστε πάρα πολύ ευαίσθητοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να μεταφέρω εδώ κάποιες σκέψεις στην Επιτροπή αυτή, γιατί πιστεύω ότι θα ήταν ενδιαφέρουσε. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στους τρεις καθηγητές για την τόσο καλή δουλειά τους, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Όντως, είναι καλό να έχουμε περισσότερες πληροφορίες, περισσότερη ενημέρωση αντικειμενική για να πάρουμε στο μέλλον αποφάσεις. Πάντως, η αλήθεια είναι, το αναγνωρίσατε κι εσείς, ότι δεν πρόκειται μόνο για μια ανάλυση κέρδους κόστους. Η πολιτική συνοχής είναι μια πολιτική αλληλεγγύης και ξεκινάμε από ένα κοινό οικοδόμημα, μια κοινή προσπάθεια που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από εκεί ξεκινάει η πολιτική συνοχής, μια πολιτική αλληλεγγύης επαναλαμβάνω. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε με άλλες πολιτικές. Η πολιτική όμως συνεργασίας και ανάπτυξης, για να πάρουμε ένα παράδειγμα. Η χώρα μου, η Ισπανία, αν και δεν πρέπει να μιλάμε εδώ για χώρες, δεν είναι και πολύ καλό αυτό, 5% προσφέρει στην πολιτική ε, συνεργασίας και ανάπτυξης. Και σίγουρα οι περισσότερε από τι χώρε που εκπροσωπούνται εδώ πέρα δίνουν πολλά για την πολιτική συνεργασία και ανάπτυξη. Εμεί έχουμε προγράμματα στη Βραζιλία, στην Κίνα, στην Αργεντινή, σε ένα μεγάλο μέρο του κόσμου δεν έχουμε τα προγράμματά μας μόνο σε χώρες που το χρειάζονται πιο επιγόντως. Εμείς έχουμε διαφοροποίησει τη σχέση μας με την ανάπτυξη και είμαστε σε πολλές χώρες. Γιατί υπάρχουν πολλές χώρες που ίσως βρίσκονται σε μια διαδικασία ανάπτυξης Παρ' όλα αυτά εξακολουθούν και να υπάρχουν προβλήματα για τα οποία πρέπει να βοηθήσουμε, γιατί πρέπει να αντιμετωπιστούν. Συνεπώς, όλες οι χώρες. Έχουμε την υποχρέωση μαζί να ορίσουμε μαζί την πολιτική συνοχή σαν μια σφαιρική πολιτική. Και αυτή η πολιτική συνοχή χρειάζεται την ελληνική όλων των χωρών, και των εισφορέων και των δικαιούχων. Και ίσως τα αποτελέσματα να μην φαίνονται τώρα, αλλά σε 10 ή 15 χρόνια θα έχουμε μια Ευρώπη με περισσότερη συνοχή εφόσον όλοι δείξουμε με αλληλεγγύη την στήριξή μας στην πολιτική αυτή συνοχής. Εμείς έχουμε εκλεγεί από τους πολίτες για να φέρουμε σε πέρα στην αποστολή να υποστηρίξουμε την πολιτική συνοχής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπάρλι, πολύ καλά υπογραμμίσατε την κατάσταση και τη σχέση Πολωνία-Ιρλανδία και είπατε γιατί η Πολωνία ως χώρα είναι στο μέσο όρο σιγά σιγά όσον αφορά το ΕΠ παρόλα αυτά ότι υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες δεν έχουν φτάσει σε αυτό το στόχο. Και αυτό που ισχύει για την Πολωνία ισχύει και για άλλες χώρες. Αναφερθήκατε και στην Ιρλανδία όπου η Νότια Ιρλανδία ε, έχει δει τον κόσμο να φεύγει προς την Ανατολική Ιρλανδία και δεν έχει ευημερίσει τόσο όσο άλλες περιφέρειες της Ιρλανδίας. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να γίνει μια επαναταξινόμηση των περιφερειών μέσα στις χώρες και σε επίπεδο κοινοβουλίου, αλλά και από την Επιτροπή άκουσα ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια τέτοια νέα επαναταξινόμηση. Εγώ όμως επανέρχομαι. Γιατί αυτό που ισχύει για την Ιρλανδία σίγουρα ισχύει και για άλλε χώρες. Ίσως είμαστε το χειρότερο παράδειγμα όπου η, η ανεργία είναι υψηλή, όπου οι δαπάνες οι δημόσιες ε, αυξάνονται, χάνονται θέσεις απασχόλησης καθημερινά και πρέπει να καταφέρει να βρει 4,5 δις η κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη χώρα Ωραία, σε πολλούς τομείς λοιπόν είμαστε στη χειρότερη κατάσταση. Και αν μάλιστα προσθέσετε σε αυτό και τα χρέη που έχει ο καθένας από εμά στην Ιρλανδία, κάτι λοιπόν πρέπει να γίνει για τις περιφέρειες όπου χάνονται συνέχεια θέσει απασχόλησης και όπου να πρόσφατα η Ντέλα έφυγε από το Λίμεριχ στην Ιρλανδία και πήγε στην Πολωνία. Ευτυχώς η Επιτροπή είπε ότι θα έπρεπε να πληρώσει γι' αυτό η εταιρεία. Πάντως όλα αυτά δείχνουν πως πρέπει να ξαναδούμε τις περιφέρειες, την κατάστασή τους. Και αν δει κανείς μια περιφέρεια, μήπως θα έπρεπε να δει και τις υποπεριφέρειες, περιοχές δηλαδή μέσα σε κάποιες περιφέρειες, γιατί μερικές φορές υπάρχουν βιομηχανικά πάρκα μέσα σε μια περιφέρεια. Βλέπετε στο Σάνον στην Ιρλανδία έχουμε μια κατάσταση. Αν πάτε προς τον Galway μπορεί να δείτε ότι δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης ενώ αν πάτε αριστερά προς το κόρτιο το Λίμερικ θα δείτε ότι η κατάσταση είναι διαφορετική και η ταξινόμηση είναι διαφορετική. Είχα συναντήσεις την προηγούμενη εβδομάδα με ομάδες από την περιοχή και ακριβώ τόνισαν ότι πρέπει να αλλάξει, πρέπει να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει και να είμαστε πιο ελαστικοί στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που προκύπτουν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης όχι μόνο στην Ιρλανδία, σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ορισμένες περιφέρειες πλήττονται πολύ περισσότερο από άλλε. Και φοβάμαι ότι αν μια χώρα σαν τη Γαλλία και τη Γερμανία ή και την Αγγλία βγούνε από την ύφεση την οικονομική, που αυτό βέβαια όλοι θέλουμε, και αν το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι τα επιτόκια αυξηθούν και πάλι, αυτό θα χειροτερέψει την κατάσταση για τους ανθρώπους και για τις περιφέρειες. Αυτό λοιπόν ήθελα να σας πω. Μήπως μπορείτε να το δείτε και να το σχολιάσετε κάπως αυτό. Ευχαριστώ. Να απαντήσει ο καθηγητής Όντιτ. Ε, äh, Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις αυτές, πολλές από τις οποίες υπερβαίνουν ε, τον στενό εστιασμό της μελέτης. Το ευρωπαϊκό έργο έχει και άλλες διαστάσεις και όχι μόνο την στενά οικονομική. Αυτό ε, νομίζω είναι αυτονόητο, συμφωνούν όλοι ότι πρόκειται για ένα θέμα συνολικά της κοινωνίας όπου βέβαια η οικονομική συνιστόσα έχει ένα ιδιαίτερο ρόλο μέσα σε αυτό το ευρύτερο σύνολο. Ωστόσο είναι σημαντική. η εφαρμογή των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών πολιτικών γίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο όπου χωρίς την ρητή συμμετοχή των νέων χωρών είχαμε μία οικονομική ολοκλήρωση. Ξεκινώντας από τις αρχές της δεκαετίας του 90, τα οικονομικά σύνορα σιγά σιγά σταδιακά καταργούνται ώστε μέχρι περίπου το 2000-2001 μπορεί να μιλήσει κανείς για την βασική αρχή μιας ζώνης ελεύθερων συναλλαγών με ορισμένους περιορισμούς. Αυτή η διαδικασία βαθαίνει με τη διεύρυνση όπου καταργούνται ορισμένα ακόμα σύνορα με την συνέπεια ότι εντελώς απροσδόκητα μετά από το 2004 υπάρχει μια σημαντική όθηση των οικονομικών εμπορικών συναλλαγών των παλαιών χωρών μελών με τις νέες. Και με, μόνο και με την απλή μείωση των, του κόστου των συναλλαγών. Και εδώ όμως ισχύει ότι η σύγκληση και η ολοκλήρωση θα γίνονταν, θα πετύχαιναν και χωρίς την Ευρωπαϊκή Διαρθρωτική Πολιτική. Πάντως ένα από τα καθήκοντά μας είναι να καταδείξουμε ποια είναι η συμβολή της Ευρωπαϊκής διαθωτικής Πολιτικής μέσα σε αυτό το πλαίσιο για την επιτάχυνση της συνοχής. Και τα συμπεράσματα της μελέτης, όπως θα είδατε, η διάκριση που γίνεται ανάμεσα στη φάση εφαρμογής και στη φάση του κόστους Αυτά τα συμπεράσματα δείχνουν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην απασχόληση και για την περίοδο μέσα στο 2000, μεταξύ 2000 και 2006. Αυτό είναι ένα τμήμα της εικόνας, αλλά σημαντικό τμήμα και αυτά γίνονται, όπως είπα, μέσα σε ένα ολοκληρωμένο οικονομικό χώρο, ο οποίος όμως βρίσκεται ακόμα σε, μέσα σε μια δυναμική παραπέρα ολοκλήρωσης. Άρα η μελέτη δεν μπορεί να φτάσει στο τέλος της με μία μόνη ανάλυση, αλλά στην πραγματικότητα βρισκόμαστε μέσα στην πορεία προς μια ακόμα περαιτέρω ολοκλήρωση μιας κοινότητας χωρών, όπου οι ευρωπαϊκές διαρθρωτικές πολιτικές πρέπει να θεωρούνται ως ένας πυλώνα, ω μια στήλη της αυτή τη ολοκλήρωση μαζί με την ε, νομισματική ένωση μαζί με τις οικονομικές πολιτικές ώστε να πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα συμπεράσματα. Και ένα τελευταίο. αναφορικά με την κατανομή των διαρθωτικών ταμείων ε, στα επιμέρους ε, υποδομές, άμεση ενισχύσει επιχειρήσεων, ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι εύκολο να λυθεί. Εξαρτάται και από το επίπεδο ανάπτυξης της κάθε κρατικής οικονομίας η οποία λαμβάνει τα κονδύλια αυτά. Έχει διαφορά τώρα Εάν για παράδειγμα η συγκεκριμένη οικονομία μάλλον αλλιώς εάν τα, τα κονδύλια διατίθενται για ε, έρευνα και ανάπτυξη σε καθυστερημένες οικονομίες ή σε ανεπτυγμένες οικονομίες. Ακόμα και αν το ανθρώπινο δυναμικό είναι ικανό και άξιο σε κάποια ε, καθυστερημένη οικονομία, υπάρχει έλλειψη υποδομών. Για να μπορέσει για να γίνει πιο επιτυχές πρέπει να μπορέσει να μετακινηθεί η καμπύλη. Και όσο περισσότερες δυνατότητες δίνεται στην έρευνα και ανάπτυξη, τόσο σημαντικότερες είναι και οι δυνατότητες ανάπτυξης ε, της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όμως, οι καθυστερημένες οικονομίες δεν θα ενισχυθούν μόνο από την έρευνα και ανάπτυξη, και όχι κυρίως, αλλά με την πιο αποτελεσματική χρήση των υφιστάμενων τεχνολογιών και με την προσθήκη και άλλων τεχνολογιών. Παράδειγμα, η αυτοκινητοβιομηχανία. Στις παλιές χώρες μέλη, η υφιστάμενη τεχνολογική γνώση μεταφέρθηκε στις νέες χώρες μέλη. Και εκεί συνδυάστηκε με τις επιτόπου με το επιτόπου εργατικό δυναμικό για να αναπτύξει νέα ανταγωνιστικότητα. Το πρώτο βήμα λοιπόν δεν είναι να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά να μεταφερθούν οι φυστάμενες τεχνολογίες που υπάρχουν στις παλαιές χώρες μέρη να μεταφερθούν στις νέες, ώστε να υπάρξει μια σταδιακή ανωδική πορεία, δηλαδή να προλάβουν οι καθυστερημένες αυτές οι οικονομίες τις άλλες ώστε να μπορέσουν μετά να προχωρήσουν και σε έρευνα και ανάπτυξη. Η δυσκολία έγκυται στο να εξευρεθούν τα κατάλληλα μέτρα και αυτά θα είναι διαφορετικά ανάλογα με την κάθε χώρα που έχει ανάγκη να ληφθούν τα μέτρα αυτά. Σας ευχαριστώ για το σχόλιο. Το λόγο θα λάβει αμέσως ο συναδελφός σας, αλλά θα δώσουμε την ευκαιρία για μία ακόμη ερώτηση από τον κύριο Τσέλερ. Äh, äh, ευχαριστώ. Με πρόλαβε λίγο ο καθηγητής Ούντιντ. Είμαι νέος ευρωβουλευτής και γι' αυτό ευχαριστώ ιδιαίτερα για την παρουσίαση. Και τώρα μέσα από την παρουσίασή σας και έχοντας ρίξει μία ματιά στο υλικό που μας διαθέσατε χαίρομαι πρώτα που επιλέχθηκε αυτή η προσέγγιση δηλαδή ενίσχυση ορισμένων πολιτικών και εν προκειμένου ε, το ποιες είναι και οι συνέπειες των διαθετικών πολιτικών και στις δωρήτριε χώρες. Δεν θα κάνω εγώ την αξιολόγηση γιατί την κάνατε ήδη. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να κάνω την πολιτική αξιολόγηση. Εξετάζοντα τώρα τα συμπεράσματά σας και ίσω λέγοντα τα κάπω υπερβολικά ή μάλλον πολύ υπερβολικά, θα πρέπει να πω τώρα στην πατρίδα μου να πω στους ψηφοφόρου ποιε είναι οι συνέπειες τη ευρωπαϊκής πολιτικής τη συνοχή τα τελευταία χρόνια και τι τελευταίε δεκαετίες. Όπως είπε και ο κ. Κορτέ προηγουμένω, για την αλληλεγγύη. Άμεση επίδραση, τουλάχιστον υπέρ των δωρητριών χωρών, αυτή ήταν απειροελάχιστη. Εκεί όπου τα χρήματα καταλήγουν μέσω της ανακατανομής από την πολιτική ε, συνοχής υπάρχουν κάποιες θετικές συνέπειες που όμως ακόμα δεν έχουν αποδείξει την βιωσιμότητά τους. Είδαμε και πριν και την παρουσίαση του ΕΣΠΟΝ που δείχνει ότι υπάρχουν περιφέρειες στην Ευρώπη που παρόλο που έχουν λάβει σημαντικά κονδύλια μέσω διαφόρων ευρωπαϊκών πολιτικών εξακολουθούν να μην μπορούν να προσεγγίσουν τον Ευρωπαϊκό Μεσόρο. Υπάρχουν άλλες περιφέρειες όπως η Πολωνία που έχουν μια ιδιαίτερη, ένα ιδιαίτερο δυναμισμό που χρειάζεται βέβαια στήριξη και με ευρωπαϊκά μέτρα που έχουν ωστόσο καταφέρει να φτάσουν σχεδόν το ευρωπαϊκό, τον ευρωπαϊκό μισόωρο. Αυτά που είπατε εσείς κύριε καθηγητά, αυτό που έχει πρώτη στη σημασία είναι να τα συνδυάσουμε αυτά, να τα εντάξουμε μέσα στην ευρύτερη ευρωπαϊκή διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μια μεμονωμένη ενατένιση της διαρθρωτικής πολιτικής, αλλά η Ευρώπη, δεν είναι απλώς μια προσπάθεια καθίδρυσης της ειρήνης, αλλά και μια ισχυρή διεθνής αγορά που να μπορεί να ανταγωνιστεί παγκόσμια. Τώρα όμως και στη βάση των, γνώσεων που δώσατε και των συστάσεων που κάνατε, αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για μένα πάντως αυτά που προκύπτουν από τις τελευταίες δύο μέρες είναι ότι η Επιτροπή μας πρέπει να κάτσει να σκεφτεί σε βάθος ποια πρέπει να είναι η μελλοντική Πολιτική συνοχής στα ευρωπαϊκά μέτρα. Νομίζω ότι έχει αρχίσει πια η συζήτηση και είμαι βέβαιος ότι θα εμβαθυνθεί αρκετά. Σας ευχαριστώ πάντως για τη συμβολή σας. Πράγματι κύριε συνάδελφε πρόκειται για πάρα πολλά χρήματα, χρήματα τα οποία αφαιρούνται βέβαια από τους προϋπολογισμούς των δωρητριών χωρών και όπου λείπουν για άλλα πράγματα. Παρακαλώ, οι συνάδελφοι, παρόλο που είναι δικαιολογημένο να ζητούν αλληλεγγύη, ας σκέφτονται και αυτοί την άλλη όψη του νομίσματος. Έχουμε δύο ακόμη ε, συνόψεις θα κάνουν οι ε, εμπειρογνώμονες. Πρώτος ο κύριος Μπράντλεϊ και τέλος ο κύριος Ζαλέσκη. Πολύ σύντομα. Ένα από τα ωφέλη για μας που συνομιλούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ότι περισσότερο έχετε ολιστική προσέγγιση εσείς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζεται στο δικό της ρόλο και μόνο. Ο πρόεδρος και ο συνάδελφος από την Ουρμανία έθεσαν το ζήτημα ότι ανοιχτό εμπόριο και άμεσες επενδύσεις είναι κινητήρια δύναμη για την, πολιτική για την συνοχή όπως και η πολιτική συνοχή. Συμφωνώ, το 1997 είχα τη δυνατότητα να συντάξω μια έκθεση τον Μάριο Μόντι όταν ετοίμαζε την αναθεώρηση της ενιαίας αγοράς με τα δεκαετία και ήθελαμε να δούμε πώς ταιριάζει η πολιτική συνοχής με την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και τα πορίσματα ήταν δραματικά οι κρατικές προμήθειες και απελευθέρωση των κρατικών προμηθειών ωφέλησαν την ε, Ιρλανδία με τα φαρμακευτικά της προϊόντα και τους υπολογιστές ενώ όλες τις χώρες συνοχής ωφελήθηκαν περισσότερο από την ενία αγορά από ό,τι ε, από, το Ταμείο Συνοχής. Έπρεπε λοιπόν να συναθρήσεις αυτά. Και ο ρόλος του Κοινοβουλίου είναι να σκέφτεται ολιστικά και να σπάσει τους φραγμούς που οδηγούν σε διαχωρισμούς και μερικές αναλύσεις. Ο κ. Κορτέζ αναφέρθηκε σε ευρύτερα θέματα για την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσης. Τα λαμβάνω υπόψη αυτά που είπε και από ό,τι κατάλαβα διατείνεται ότι θα έπρεπε να, σκεφ... να δούμε την πολιτική, την ευρωπαϊκή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσης στα ίδια πλαίσια με το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τρίτο κόσμο. Και αν τα δείτε όλα αυτά ενιαία, θα δείτε πιο θετικά την πολιτική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσης και πώς λειτουργεί στην Ευρώπη. Δεν θα θεωρηθεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια σε τρίτες χώρες είναι μια σπατάλη διότι δεν υπάρχει συνεργασία με τις κυβερνήσεις όπως γίνεται εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και γίνεται μια απεμπόληση και όσον αφορά τα χρήματα. Και αν δίνετε τους πόρους που διατίθεται όσον αφορά τη συνοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πολύ περισσότερα από ό,τι δίνονται στις ε, προσαχάριες χώρες της, ε, Ευρω... Αφρικής. Ε, αυτά θα πρέπει να τα λαμβάνει υπόψη το Κοινοβούλιο και τα μαθήματα που βγαίνουν από την πολιτική συνοχής και τα σφάλματα που έγιναν και οι σπατάλες που έγιναν, όλα αυτά θα πρέπει να τροφοδοτούν τη συζήτηση σχετικά με το ρόλο της Ευρώπης αναπτυξιακή πολιτική στις πραγματικά φτωχές χώρες. Και τέλος, ο Ιρλανδός συνάδελφος αναφέρθηκε στα, στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες και θα μπορούσα ειλικρινά να απαντήσω εφόσον είναι Ιρλανδός πιο ελεύθερα θα το απαντήσω εφόσον συμπατριώτησα από ό,τι απαντούσα σε κάποια άλλη χώρα. Στην Ιρλανδία είδαμε ότι είναι μια διαδοχική διαδικασία η περιφερειακή ανάπτυξη. Πρέπει να δώσει προτεραιότητα σε κάποιε περιφέρειες για να προωθηθεί η ανάπτυξη και τραβάνε πίσω του αυτέ οι περιφερειε, άλλε περιφέρειε Δεν είναι αυτόματη διαδικασία, χρειάζεται έξυπνη αντιμετώπιση ε, για να λειτουργήσει χωροταξική αλλά και ακόμα και αρνητικέ δυνάμει και ε, η κυκλοφοριακή συμφόρηση σε πόλεις ε, οδηγούν τη βιομηχανία σε άλλες περιοχές όπως πάνε και εταιρείε σε περιφερειακές χώρες για την παραγωγή των προϊόντων τους. Δεν θα πρέπει να αντιδρούμε όταν υπάρχει κρίση και να ζητάμε μεταφορά πόρων προς τις περιοχές. Τότε, σαν μόνη λύση για να βοηθηθούν οι περιφέρειες που υποφέρουν, Πρέπει να δείτε πώς λειτουργούν οι χώρες, τι μηχανισμούς έχουν, όπως η Πολωνία και οι πλουσιότερες περιοχές της Δύσης που μαγνητίζουν και τραβούν τις ανατολικές περιοχές και δίνουμε στην ευκαιρία στις ανατολικές περιοχές να εφαρμόσουν άλλη πολιτική συνοχή. Αντί να φτιάχνουμε στην Ανατολική Πολωνία εργοστάσια και αυτοκινητοδρόμους και κοντά στην Ουκρανία, καλύτερα να εξασφαλίσουμε το να χρησιμοποιούν τι ευκαιρίε που έχουν πλήρω οι δυτικέ περιοχές. Και εσωτερική αλληλεγγύη όμω χώρας πρέπει να διατηρηθεί. Η διαδικασία περιφερειακή οροπία είναι κάτι πολύ φίνο. Και αν υποστηρίζονται περισσότερο κάποιε περιφέρειε από άλλε, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι αποτυχία τη πολιτική συνοχή. Ε, Σα ευχαριστώ. Τελειώνει ο κ. Ευχαριστώ πολύ. Τα κράτη τα οποία χρηματοδοτούν την πολιτική συνοχή μπορούν να έχουν κάποια κέρδη. Φυσικά είναι συζητήσιμο. Φτάνει, είναι πολύ, είναι λίγο. Όμως πιστεύω ότι η ανάλυση μας έχει δείξει ότι τέτοια πλεονεκτήματα υπάρχουν για τις χώρες εισφορής. Βέβαια, η συνοχή δεν είναι μόνο οικονομική απόδοση. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε μια άλλη διάσταση. Η πολιτική συνοχή είναι μια πολύ πρακτική μέθοδος προκειμένου να φτιάξουμε μια αποτελεσματική δίκηση στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες που βρίσκονται κάπως πίσω, ιδιαίτερα στις νέες χώρες μέλη. Ακριβώς λοιπόν, η δίκηση πρέπει να είναι αποτελεσματική. Γιατί εκείνη είναι που φροντίζει ώστε οι διάφοροι κανόνες, οι ευρωπαϊκές διατάξεις, οι νόμοι να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο παντού. Αν η δίκηση δεν είναι αποτελεσματική, τότε οι οδηγίες δεν θα εφαρμόζονται καλά και η πολιτική συνοχής μεταξύ άλλων δεν θα προχωρήσει όπως πρέπει. Μιλήσαμε κάπως για την μετεγκατάσταση, για την Ντέλ που έφυγε από την Ιρλανδία για παράδειγμα και που βρίσκεται σήμερα στην Πολωνία, στην πόλη Λότς. Υπήρξαν και άλλες μετεγκαταστάσεις όμως. Η φαντουργία στην ε, Πολωνία και τώρα φύγανε και από την Πολωνία και πήγαν ακόμα πιο μακριά, στην Ουκρανία ή στη Μολδαβία φυσικά δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη βιομηχανική παραγωγή στην Ευρώπη. Πρέπει να φροντίσουμε να την κρατήσουμε στην Ευρώπη, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνο από υπηρεσίες. Η μετεγκατάσταση λοιπόν μέσα στην Ευρώπη είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποτελέσει πλονέκτημα για όλους μας. Μην νομίζουμε ότι το σύνολο των κερδών πηγαίνει στις χώρες όπου εγκαθίσταται τελικά η παραγωγή. Το βασικό για μας είναι η παραγωγή να μην φεύγει από την Ευρώπη. Αυτό θα ήταν μεγάλη απώλεια για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Είναι μια συζήτηση πολύ ενδιαφέρουσα βέβαια αυτή, η οποία μας επιτρέπει να ρίξουμε λίγο φως στην πολιτική συνοχή στις μέρες μας. Μιλήσαμε για τα θετικά της πολιτικής συνοχής στις πιο καθυστερημένες οικονομικά περιοχές της Ευρώπης. Μιλήσαμε και για τις θετικές πτυχές της συνοχής και στις χώρες εισφορής. Εμένα μου άρεσε αυτό που είπε ο κύριος Μπράτλεϊ, ότι οι χώρες εισφορής εποφελούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την εσωτερική αγορά. Τα τελευταία χρόνια η Γερμανία είχε ε, πλεονέκτημα πάνω από 5 δις ευρώ. Κατά συνέπεια λοιπόν είναι υποχρέωσή μας την αλληλεγγύη να την εφαρμόζουμε. Αυτό που μάθαμε σήμερα είναι ότι τελικά χάρη στην πολιτική συνοχή μπορούμε να έχουμε μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Είναι δυνατόν αυτό αλλά βέβαια σε ορισμένου τομεί πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, ώστε αυτή η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία να ε, βοηθήσει κάποιες περιφέρειες και ώστε να γίνει ακόμα πιο δυνατή στις ορισμένες χώρες της φορής. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τις εμπειρογνώμονες για τα όσα μας είπανε. Ευχαριστώ επίσης για την προετοιμασία της συνεδρίασης αυτής και απλώς και μόνο έχω να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίαση προβλέπεται στις 2 Δεκεμβρίου 3 με 6,5 και μετά 3 Δεκεμβρίου 9 με 12.